Μπορούμε να αρχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αρχίζουμε λοιπόν σήμερα το πρωί πρώτα απ' όλα με την έγκριση της ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σα πω το εξή. Τώρα, σε σχέση με την ημερήσια διάταξη την οποία έχετε λάβει, πρέπει να πω ότι η κυρία Λουβά μα ζήτησε το σημείο 5 για το χέλι να το συζητήσουμε τον Ιανουάριο. Το σημείο 7 τη συμφωνία με την Μαυριτανία. Η Κομισιόν ζήτησε αν είναι δυνατόν να το συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα. Άρα θα το εξετάσουμε αμέσως μετά την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Ντεκούχτ. Μετά το 9. Λοιπόν, θα περάσουμε στο 7. Και μετά από το σημείο 8 θα μπορούσαμε να ε, έχουμε ένα νέο σημείο 8α για να συζητήσουμε τις διαπραγματεύσεις με την ΙΚΑΤ και τα αποτελέσματα. Εάν συμφωνείτε, περνάω σε ανακοινώσει του Προέδρου, δεν έχω από τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα καινούριο, άρα περνούμε αμέσως στη σημείο 3 την τροποποίηση του κανονισμού 1098-2007 του Συμβουλίου τη 18 Σεπτεμβρίου τη Σύσταση Πολιτού Σχεδίου του αποθέματα γάλα στην Βαλτική τη Αλευτική Δραστηριότητα που εκμεταλλεύονται αυτά τα αποθέματα. Έχουμε ψηφοφορία. Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ε, αν έχει όλα καλώς, θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για να πάμε πιο γρήγορα. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Δεν έχω, κάρτα, δεν έχω κάρτα για την ψηφοφορία. Εντάξει, θα μετρήσουμε ε, την ε, <coughs> ψήφο σας. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν άρα προβλήματα. Θα δώσουμε χρόνο στην κυρία Τόμας να βγάλει την κάρτα της και θα αρχίσουμε. Λοιπόν, περνάμε αμέσως στην ψηφοφορία. Τροπολογία 23. Αρχίζει η ψηφοφορία, κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία αριθμός 1. Αρχίζει η ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ε, περιμένω. Ξαναρχίζουμε, λέει ο πρόεδρος. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. και ο κύριος ε, Σαλαβράκος δεν έχει την κάρτα του, θα μέτρηθει η ψηφοφορία. Θα θέλαμε να έχουμε τα αποτελέσματα της ε, ψηφοφορίας στην ε, οθόνη, παρακαλώ. Λέει η κυρία Λεβίν. Ε, αν δεν κάνω λάθος, λέει ο πρόεδρος, στην συμβαστική τροπολογία 2 υπήρχαν τέσσερι αντίθετοι ψήφοι και δύο αποχές. Τροπολογία 6. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται συν ε, δύο ψήφους που μετρήσαμε από συναδέλφους που δεν έχουν την ηλεκτρονική τους κάρτα, λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 29. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 8. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 9. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη. Ποιος είχε σηκώσει το χέρι για να ψηφίσει παρακαλώ για να γίνει η καταμέτρηση υπέρ και κατά, άρα εγκρίνεται. Λοιπόν, θα ξαναψηφίσουμε, αλλά να είμαστε σαφείς. Όποιοι δεν έχουν την κάρτα, να αφήσουν το χέρι σηκωμένο για να μετρήσουμε. Λοιπόν, Ξαναψηφίζουμε την τροπολογία 9. Αρχίζει η ψηφοφορία. Υπέρ. 11 προς έντεκα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 30. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Συγγνώμη, αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 13. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 14. Αρχίζει, λίγη, εγκρίνεται. 15. Αρχίζει, λίγη, εγκρίνεται. 16. Αρχίζει, κλείνει, εγκρίνεται. 17 αρχίζει, λίγη, εγκρίνεται. 18. Αρχίζει, λίγη, εγκρίνεται. 1. Αρχίζει, λίγη, εγκρίνεται. 19. Αρχίζει, λίγη, εγκρίνεται. 20 που αντικαθιστά την 2. Αρχίζει, λίγη, εγκρίνεται. 21, αρχίζει, λίγη, εγκρίνεται. 3, αρχίζει, λίγη, εγκρίνεται. 22, αρχίζει, λίγη, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την νομοθετική πρόταση έτσι όπως την τροπολογήσαμε. Αρχίζει, λίγη, εγκρίνεται και το σύνολο της, του νομοθετικού ψηφίσματος αρχίζει, λίγη, εγκρίνεται με 15 προς 4 και μία αποχή. Το ψήφισμα. Κύριε Βαλέσσα, συγχαρητήρια. Περνούμε τώρα στο επόμενο σημείο, που είναι η τροποποίηση του κανονισμού 812-2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεπίπτοντα αλλιεύματα κοιτοειδών κατά την αλληλεία και για τροποποίηση του κανονισμού 88 Παύλα 98. Αν θυμάστε, στις 8 Οκτωβρίου μας παρουσίασε την πρότασή της η Επιτροπή και σήμερα θα έχουμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Η είναι ο κύριος Ρόμεβα. Του δίνω μέσο στο λόγο. Κύριε Ρόμεβα, έχετε μέσο στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω να έχει ησυχία στην αίθουσα. Καλημέρα σας. Πρόκειται για ένα τεχνικού περιεχομένου θέμα σε σχέση με την πρόταση λισαβονοποίησης. Περιμένω, περιμένω, περιμένω πρόεδρε να ηρεμήσει το σύνολο των συναδέλφων για να μπορέσω να συνεχίσω, λέει ο κύριος Ρωμέβα. Ησυχία, ηρεμία, σιωπήστε, λέει ο πρόεδρο. Συνεχίζω. Λοιπόν, θα είναι πολύ σύντομο το θέμα αυτό, διότι πρέπει να πω ότι εδώ πρόκειται για λισαβονοποίηση του κανονισμού που αφορά τα κοιτοειδή. Είχα κάποιες επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από όσον κατάλαβα, και εγώ Διάβασα τον κανονισμό 88-98, στον οποίο πρέπει να γίνει αυτή η μικρή τροποποίηση. Μόνο ένα μικρό σημείο είναι αυτό το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε. Σε σχέση με το άρθρο 1, βασικά με τα ε, εξοπλισμό που αφορά την, ε, τον ήχο τις συσκευές, δηλαδή τις αποτρεπτικέ ακουστικές συσκευές συγκεκριμένα. Η σύστασή μου είναι να ακολουθήσουμε την πρόταση της Επιτροπής χωρίς να προσθέσουμε τίποτε περαιτέρω. Ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα. Κύριε Αρσένη. Thank you, President. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε ο συνάδελφος, ο κύριος Ρωμέδα είναι πάρα πολύ τεχνική η έκθεση. Είναι όμως μια ευκαιρία για να συζητήσουμε το θέμα των κοιτοειδών, διότι είναι προβληματικό. Και πώς θα διαχειριστούμε τα αποθέματα των κοιτοειδών εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αντίθετα με τις ε, όπου υπάρχει σχετική νομοθεσία για τα θαλάσσια κοιτοειδή, εδώ δεν υπάρχει νομοθεσία για την προστασία των θαλασσίων ε, κοιτοειδών. Και νομίζω ότι είναι κατάλληλη ώρα τώρα να ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει πρόταση γενικότερα για τα θαλάσσια θηλαστικά και ειδικότερα για τα κοιτοειδή διότι έχουμε αποσπασματικά νομοθετήματα, αλλά όχι μια σφαιρική νομοθεσία που να ενέχει όλα τα επιμέρους στοιχεία, εξασφαλίζοντας έτσι τον κατάλληλο έλεγχο και παρακολούθηση. Οπότε πιστεύω ότι είναι κατάλληλη ευκαιρία για να το συζητήσουμε. Ευχαριστούμε κύριο Στίβενσον. Τώρα ευχαριστώ, Πρόεδρε αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για μια τεχνική έκθεση νομικής φύσεως, αλλά δράτουμε τις ευκαιρίες για να θέσω μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από ό,τι καταλαβαίνω, μου λένε πολλοί αλληλείς ότι δεν λειτουργούν σωστά αυτές οι αποτρεπτικές ακουστικές συσκευές ε, και ενίοτε έχουν και τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ε, τα κοιτοειδή εξοικειώνονται με τον ήχο που εκπέμπουν αυτές οι ακουστικές ε, συσκευές και θεωρούν ότι είναι πηγή τροφής και άρα έλκονται από, τα, από τις συσκευές αυτές. Ε, λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος ακριβώς ε, της νομοθεσίας αυτής. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, απαντήσει. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κανένας άλλος ε, που ζητάει το λόγο. Όχι, τότε ο κύριος Μπιάνκι από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρωμέβα για την υποστήριξη του, για την τεχνική πτυχή αυτή της πρότασης και της κατεξοδότησης πράξης που προτείνουμε για το άρθρο 31 τα σημεία που αναφέρει ο κύριος Αρσένης και ο κύριος Στίβενσον θα σκεφτώ το αίτημα σας να προβληματιστούμε για ένα γενικότερο κανονισμό πλαίσιο για την προστασία των κοιτοειδών. Είχαμε την ευκαιρία, αν δεν κάνω λάθος, να εξηγήσουμε όταν παρουσιάσαμε τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής ε, πολιτικής ότι η πρόθεσή μας είναι να κοιτάξουμε με κριτικό πνευμα τι έχουμε στο πλαίσιο του ε, νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων που θα λάβουμε αμέσως μετά από τη μεταρρύθμιση ώστε να εκαθαρίσουμε κατά κάποιο τρόπο και να δημιουργήσουμε συνοχή, ένα συνεκτικό σύνολο κανόνων για τις καθημερινές δραστηριότητες των αλλιέων αντί να δημιουργήσουμε ένα συγκεκριμένο νόμο. Θα εξετάσουμε το έτοιμά σα και θα επανέλθει η Κομισιόν σε εσά με αυτό. Τώρα το ζήτημα που αναφέρει ο κ. Στίβενσον για τι ακουστικέ συσκευέ ε, αληθεύει σε ορισμένες περιπτώσεις έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και πάλι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σκοπεύουμε να μελετήσουμε στο προτινόμενο αναθεωρημένο πλαίσιο τεχνικών μέτρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλε παρεμβάσει. Ο κύριο Ρόμεβα. Για να απαντήσω, και εγώ το ίδιο θα έλεγα, όπω η Κομίσια, όντω, τα δύο θέματα τα οποία έθεσαν οι συνάδελφοι, κυρίω η παρατήρηση του κυρίου ε, Αρσένη είναι κάτι το οποίο και εγώ θέλω να πω, αλλά νομίζω ότι με την πρώτη επιτροπή νομίζω ότι μέσα σε ευρύτερο πλαίσιο θα χειριστούμε το θέμα. Πολύ πιο συγκεκριμένα από ότι τώρα για αυτή την συγκεκριμένο κανονισμό. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, προθεσμία Κατάθεση τροπολογικό σημείο Ιανουαρίου, ψηφοφορία το Φεβρουάριο. Περνούμε τώρα στο σημείο 6, σύσταση. Μακροπρόθεσμο σχεδίο για τα αποθέματα γάδου και τι ελευτικέ δραστηριότητε που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα. Αυτό, όπω ξέρετε, πρόκειται για το δεύτερη ε, πρόταση. Η πρώτη πρόταση για την οποία επίσης ήταν η κυρία Ντόντς, ήταν κάτι που συζητήσαμε. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, 6 Νοεμβρίου, μας παρουσίασε την ε, πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σήμερα θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτή την ε, έκθεση. Δίνω αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Ντόντς. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Διάβαζα και πάλι ε, την παρουσίαση που ήθελα να σας κάνω σήμερα το πρωί. Γι' αυτό καθυστέρησα. Με ιδιαίτερη προσοχή. Την περασμένη εβδομάδα έκανα πολλές διαβουλεύσεις και από την τελευταία μας συνεδρίαση που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο που μετήχα στις συζητήσεις των συντονιστών για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Εξέτασα το θέμα λοιπόν και ζητώ συγγνώμη διότι σε αυτό το στάδιο είναι κάπως μακροσκελής η παρουσίασή μου. Τις περασμένες ημέρες μου εδόθη η ευκαιρία να συζητήσω με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΙ, με την, ε, το γραφείο της Επιτρόπου Δαμανάκη, με αξιωματούχους ε, της Ιρλανδίας του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσώπους ε, του κλάδου και φυσικά συναδέλφους βουλευτές. Θα συναντηθώ κατηδίαν με την Επίτροπο Δαμανάκη σήμερα για αυτό ακριβώς το θέμα. Την περασμένη Παρασκευή διοργάνωσα στην εκλογική μου περιφέρεια ένα πρόγευμα όπου ο Υπουργό Γεωργία Αλία και πρώην ε, βουλευτή του Κοινοβουλίου Σάιμον Κόβνη ήταν ε, επίτιμο καλεσμένο και μεταξύ των ερωτημάτων που του έθουσε είναι το εξή. Εφόσον η Ιρλανδία θα αναλάβει την Προεδρία την 1η Ιανουαρίου, ποιε είναι οι προθέσει του τόσο ώστε να δώσει μία απάντηση στις συγκρούσεις αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση με άμεση αναφορά στη μεταρρύθμιση κοινή ελευτικής πολιτικής και το μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης των αποθεμάτων κάδο. Ο κύριος Κόβνη μου υπενθύμησε σε μένα και στους υπολοιπούς προσκεκλημένους ότι ε, η δουλειά του είναι να προωθεί τα θέματα του χαρτοφυλακίου του. αυτό ισχύει και για ε, και για Εθνικού εθνικούς βουλευτές ε, και όντω χρειάζεται πρόοδος ε, στον τομέα της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Ε, για το μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης γάδου έχει κέρια σημασία κατά τη γνώμη το 2011 έγινε αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων σχεδίων διαχείρισης και η Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή κατέληξε στα εξή συμπεράσματα ότι δεν λειτουργεί σωστά το σχέδιο διαχείρισης και δεν έχει την στήριξη των εμπλεκομένων σε διάφορες περιοχές Χρειάζεται όμως αυτή η υποστήριξη για να στεφτεί με επιτυχία το μακροπρόθεσμο αυτό σχέδιο διαχείρισης. Ε, κατόπιν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χρειάστηκε 14 ολόκληρους μήνες για να καταθέσει σχέδιο μεταρρύθμισης του μακροπρόθεσμου σχέδιου διαχείρισης. Ε, με προσοχή το καλωσορίζουμε και ε, θέλουμε εγώ και όλοι οι εμπλεκόμενοι να συμβάλλουμε στην διαδικασία. Τις ε, περασμένες εβδομάδες ε, θα να μάλλον απογοητευμένοι διότι ούτως ή άλλως έχουμε καθυστερήσει και κολλησιεργεί ακόμη περισσότερο το Συμβούλιο. Ε, συγγνώμη Πρόεδρε, αλλά δεν μπορώ να συγκεντρωθώ με όλες τις συζητήσεις και τα πηγαδάκια μέσα στην αίθουσα είναι κέρια ζωτική σημασία στο θέμα για την Επιτροπή μας και πιστεύω ότι θα πρέπει το προσωπικό να ε, το σεβαστεί αυτό και να μην κάνει φασάρια. Λοιπόν, 14 μήνες αναμονής για να λάβουμε το, την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και τώρα ε, ε, το Συμβούλιο θα αρχίσει να τροποποιεί αυτή την, για να λιώνει αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, κίνημα που υποστηρίζουν διάφορα κράτη-μέλη. Στην ομάδα εργασίας ε, του Συμβουλίου η Γαλλία πρότεινε κάποιες επιτυχές ε, της μεταρρύθμισης να αλλάξουν διότι δεν συνάδουν με το άρθρο 43 της Συνθήκης Λισαβόνας του τεστ είναι, δεν εμπίπτουν στη διαδικασία συναπόφαση. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στο άρθρο 9 σε σχέση με τον προσδιορισμό των ΤΑΚ και το άρθρο 11 για τι αλλιευτικέ προσπάθειε Πρότεινα να αφαιρεθούν από το τροποποιητικό σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανταυτού να υπαχθούν σε μια νέα πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου αυτή τη φορά. Αντιλαμβάνομαι ότι η πρόταση θα συζητηθεί περαιτέρω και θα ψηφιστεί στα τέλη τη εβδομάδα σε επίπεδο κορεπέρ. Χρειάζεται όμω ομόφωνο σύμφωνη στήριξη από πλευρά των κρατών μελών για να εγκριθεί η πρόταση και βάσει των πληροφοριών που έχω όμω είναι εφικτό, είναι, είναι πιθανή μια τέτοια έκβαση. Να εξηγήσουμε τώρα γιατί το επιδιώκει αυτό το Συμβούλιο. Υπάρχει το θεμελιώδε ζήτημα των αρμοδιοτήτων για το θέμα αυτό. Για κάποιου ο στόχο είναι να ε, εξασφαλίσουμε πάγωμα των αλληλευτικών προσπαθειών, δηλαδή να μείνουμε στο 2000, ε, ε, στα επίπεδα 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, θα ε, καταθέσει τροπολογίες που θα οδηγήσουν σε πάγωμα στα επίπεδα το 2013. Εγώ υποστηρίζω το πάγωμα των αλλιευτικών προσπαθειών. Θεωρώ όμως για την ανάκτηση του αποθέματος και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας ε, της προσπάθειας του αλλιευτικού στόλου κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Βάσει της έκθεσης Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής ε, δεν είναι πολύ πιθανό ότι η μειώση των αλλιευτικών προσπαθειών ε, θα οδηγήσουν ανάλογα και σε μείωση της εθνισιμότητας των ψαριών. Οι περιορισμοί των αλλιευτικών προσπαθειών είναι βασική ατέλεια του μακροπρόθεσμου σχέδιου διαχείρισης. Τέλος της παράθεσης. Ε, εγώ φοβάμαι το εξή, παρότι υποστηρίζω το πάγωμα. Ακολουθώντας αυτήν την οδό, ελοχεύει ο κίνδυνο να θέσουμε εν κινδύνο άλλα επιμέρου στοιχεία τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τα οποία θα σχολιάσω κατά τη διάρκεια τη παρουσίασή μου. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ στην Επιτροπή, σε αυτό το χρονικό στάδιο, ότι το Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει αδίποτε θέση σε σχέση με την, ε, τη διχοτόμηση του κανονισμού Γι' αυτό και είναι πρόωρο ε, είτε για το Συμβούλιο είτε για το Κοινοβούλιο να αποταθούν ε, προ γνωμοδότηση στο δικαστήριο σε σχέση με τι αρμοδιότητε ε, και τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 9 και 11. Εάν όμω υποχρεωθούμε να ακολουθήσουμε αυτήν την άγουσα, πέραν κάθε αμφιβολία, θα περιπλακεί περισσότερο μία σειρά ζητημάτων για τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείριση πολλαπλών ειδών και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσει συνολικά για τη μεταρρύθμιση κοινή πολιτική. πολιτικής. Ε, φυσικά δεν με ικανοποιεί αυτή η προοπτική και σίγουρα θα συμπαραταχθείτε κι εσείς. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε αυτήν την εξέλιξη. Ε, αυτό ισχύει για τα αποθέματα του γάδου και για την θέση της βιομηχανίας και μην ξεχνάτε, όταν ακολουθήσουμε αυτήν την οδό θα έχουμε και άλλες παράπλευρες αρνητικές επιπτώσεις. Ακόμη και σε αυτό το στάδιο ζητώ από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να επιδιώξουν την εξέβρεση ε, εναλλακτική συμβαστική λύση. Ε, Πάντω, ε, εγώ θα ήθελα να συνεχίσω να προωθώ αυτήν την έκθεση στο όνομα τη Επιτροπή. Ελπίζω να τα καταφέρουμε καλύτερα. Το Δεκέμβριο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μέσω κανονισμού του Συμβουλίου πάγωμα των αλλιευτικών προσπαθειών. Αλλά αυτό είναι βραχυπρόθεσμο μέτρο και για κατανάλωση από τον τύπο. Αλλά τι μπορεί κανεί να περιμένει μέσω μακροπρόθεσμα. Στο επεξηγηματικό σημείωμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στο ότι αυτό συνιστά ενδιάμεση λύση, διότι αναμένουμε το πολιετέ σχέδιο δύο πολλαπλών ειδών βάσει τη μεταρρύθμιση κοινή αλλιευτική πολιτική για τη Βαλτική και για τη Βόρεια Θάλασσα. Αυτό έχει σχεδόν γίνει, αλλά για την Ιρλανδία και την Δυτική Σκοτία δεν έχουν προχωρήσει. Όντω έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά χρειαζόμαστε ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για τι εξελίξει και για να καλύψουμε τι γκρίζε ζώνε, ε, ε, ε, οι οποίε οφείλονται σε έλλειψη επιστημονικών στοιχείων και ξέρω ότι ε, αυτό δημιουργεί προβλήματα και στο σχέδιο για τη Βαλτική. Το προτινόμενο, η προτινόμενη μετατροποποίηση του άρθρου 11 και μπαίνω τώρα στα επιμέρου σημεία του ε, σχεδίου έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την ε, χρήση αποφυγής μαλίευσης του γάδου. Πολύ ωραία, αλλά χρειαζόμαστε και κάτι περισσότερο για την κατανομή των περιοχών, το είδος των δικτυών και επίσης τα 350 μέτρα της περιμένουμε τον επιλεκτικό μηχανισμό και επίσης ε, τις διάφορες διαφορετικές ανάγκες που έχουμε ανά εποχή. Το άρθρο 6 επιδιώκει να αποκλείσει τα ε, σκάφη που δεν έχουν πλήρως τεκμηριωμένη αλία από το πεδίο εφαρμογής ε, του κανονισμού Πρέπει να μεριμνήσουμε τόσο ώστε να εφαρμοστεί σωστά αυτή η διάταξη και το άρθρο 4, 4, πρέπει να διαγραφεί. Άρθρο 13, εδάφιο 2, υποσημείο Β. Εκεί διευκρινίζουμε την ερμηνεία ε, της, ε, του κανόνα σύνθεσης για το γάδο ε, στα έξω του 5% γιατί θα πρέπει να συνδυαστεί με την περίοδο διαχείριση ε, και όχι να αποφασίζεται κατά περίπτωση, αλλιώς θα αυξηθούν οι απορρίψει του γάδου. Αυτό πρέπει να το καλωσορίσουμε. Τέλος, ε, τα κράτη-μέλη σίγουρα θα επιθυμούν διευκρίνηση σε σχέση με τις πρόσθετες απαιτήσει ε, που προγραμματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει τώρα 14 του κανονισμού αυτού. Πρόεδρε, αυτό σας δίνει μια πρόγευση των ε, τροπολογιών με τις οποίες, θέλω να, τις οποίες μάλλον θέλω να επεξεργαστώ σε συνεργασία με τους συναδέλφους και ευελπιστώ ότι με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας θα μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά και όπως είπε η Επιστημονική, Οικονομική και Τεχνική Επιτροπή χρειάζεται οπωσδήποτε υποστήριξη από του εμπλεκόμενου φορεί για να πετύχουν τα μακροπρόθεσμα σχέδια. Ε, καλό το Συμβούλιο να μην ακολουθήσει αυτή την οδό. Είναι σημαντικό το πάγωμα των αλληλευτικών προσπαθειών, αλλά αν κολυσιεργήσει και άλλε εβδομάδε το Συμβούλιο θα είναι μεγάλο το κόστο, ε, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η προσπάθειά μα πριν λήξει η θητεία μα. Ε, ε, θα ήθελα λοιπόν, απευθυνόμενη στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, να τονίσω ότι είναι μια κρίσιμη καμπή ε, και για τις σχέσεις μας με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και το πώς καταφέρουμε να κινηθούμε ως Επιτροπή Αλίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ντότσο. Κύριος Καντέκ. Ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Μερικές παρατηρήσεις πρώτα απ' όλα. Τα άρθρα 12 και 13 όπως έχουν τροποποιηθεί δεν ακούγονται τα αγγλικά. Μια στιγμή παρακαλούμε. Ακούγονται τα αγγλικά. Δεν ακούγονται τα αγγλικά. Ακούγονται τώρα. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ τον Πρόεδρο ξανά που μου δίνει το λόγο και ευχαριστώ και πάλι την Διάν για την παρουσίασή της. Λοιπόν, για τρίτη συνεχή φορά. Ευχαριστώ ξανά. Et je vais remercier Diane pour sa présentation. Ευχαριστώ λοιπόν την Διάν για την παρουσίασή τη. Κάποιε παρατηρήσει Τα άρθρα 12 και 13 όπω τροποποιήθηκαν οι είναι συμβατά με τη μείωση αλληλευτικών προσπαθειών που επιθυμεί τόσο ο τομέας όσο και η Κομισιόν. Παραμένουν κάποια προβλήματα με το άρθρο 4 όσον αφορά το ε, νομιόμορφο υπολογισμό των προσπαθειών. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την τρέχοντα υπολογισμό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να απλουστεύσουμε το σύστημα Ωστόσο η τεκμηρίωση, η απαραίτητη τεκμηρίωση που αποδεικνύει ότι ε, τηρούμε αυτά τα κριτήρια ε, δεν είναι απαραίτητα πιο απλή. Η έννοια των περιοχών, για παράδειγμα, του μπακαλιάρου. Επιπλέον εισάγεται η έννοια της εξαίρεσης ε, ανα περιοχή το άρθρο 11 γάμα που εξαιρεί τα σκάφη που ε, συμμετέχουν σε πειραματισμούς ποσοστώσεων ε, αλλιευμάτων πρέπει να διευκρινιστούν κατά την άποψή μου ώστε να πλησιώνουν σωστά αυτούς τους πειραματισμούς το τροποποιημένο κείμενο του αρθρού 14 απαλά στα κρατημέλια την υποχρέωση λήψης μέτρων όταν ε, κάποια αλλιεύματα προσφέρουν υψηλό ποσοστό. Καλό είναι αυτό, Αντιθέτως δεν θα ήταν σωστό να χρησιμοποιηθεί αυτή η έκθεση, αυτό φοβάμαι, όπως και την έκθεση για τη διαχείριση του Σκάγκερακ, ώστε να επιβληθεί μια υποχρέωση ε, εκφόρτωσης. Το λέω εδώ, διότι αυτή η έκθεση αφορά ε, όλα τα αποθέματα μπακαλιάρου και του Σκάγκερακ. Όπως φαίνεται και κατά μια περίεργη συγκυρία, η πριν ακριβώς από την ψηφοφορία για το βασικό έγγραφο, η Νορβηγία δεν δέχεται ε, ε, τη διαχείριση, αποθεμα... τη απορρίψεων και μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό ότι η Νορβηγία ξαφνικά κάνει ενό είδου επανάσταση, ενώ εδώ και 30 χρόνια έχει ε, επιβάλει υποχρέωση απόρριψη, εκφόρτωσης. Και τη στιγμή ακριβώς της πρότασης αυτής ε, ε, ε, εμείς θέλουμε να εφαρμόζουμε φυσικά τους ίδιους κανόνες και σε εμά και στους γείτονες. Ίσως να είναι τυχαίο, αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω, το γνωρίζετε όλοι, ότι παρότι είμαι υπέρ της σημαντικής μέγιστης δυνατής μείωσης των απορρίψεων, θα ήθελα τα κρατημέλη να λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να μειώνουν σημαντικά τα ανεπιθύμητα αλλιεύματα. Αλλά όχι πέραν αυτού, διότι μου φαίνεται αδύνατο. Ε, ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριο Στίβενσον, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα απ' όλα την Νταϊάν Ντότς για τις διεξοδικές διαβουλεύσεις που έκανε, διότι ε, πραγματικά ε, βρέθηκε μέσα σε ένα δίχτυ και κυκλωτικό και τράβηξε το σχοινάκι το Συμβούλιο και έχει κλειστεί μέσα σε αυτό το δίχτυ. Ε, πρόκειται ε, για, ένα, για πολύ περίπλοκες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα τα τελευταία τέσσερα χρόνια με την έκθεση του Πάτε Κόμπ Γκάλαχερ, τη δική μου, ε, Μπίσκι, πάρα πολλές εκθέσεις. Ε, που κρατά στο, σε ομοιρία στην πρώτη ανάγνωση το Συμβούλιο και τώρα έγινε μια νέα εντυπωσιακή κίνηση από πλευρά του Συμβουλίου. Λέει η κυρία Αντό ότι θα διαγράψει το άρθρο 9 και 11 και τα ΤΑΚ το Συμβούλιο, να το αφαιρέσουν δηλαδή από την έκθεση και να το παραπέμψουν στην επόμενη στο επόμενο Συμβούλιο Αλίας. Ε, αυτό είναι κόλαφος ε, για την εργασία που γίνεται εδώ στο Κοινοβούλιο και μπορώ να σας πω ότι μετά το Συμβούλιο του Ιουνίου ε, δείπνησα στις Βρυξέλλες με τον Υπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και τους τρεις περιφερειακούς υπουργούς από το Ηνωμένο Βασίλειο και όταν ήγηρε αυτό το ζήτημα της εμπλοκής στο Συμβούλιο για τα μακροπρόθεσμα σχέδια οι υπουργοί κουνούσαν ε, απονενοημένα το κεφάλι τους και κοιτούσαν τους αξιωματούχους, υψηλούς αξιωματούχους που ήταν εκεί, ε, αναρωτώμενοι τι συμβαίνει. Ούτε οι υπουργοί δεν ξέρουν και μόνο οι ε, ανώτατοι αξιωματούχοι στις ομάδες εργασίας ε, γνωρίζουν τι γίνεται και θέλουν να διατηρήσουν την εξουσία για αυτό η κοινωνική υπηρεσία ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα ακόμη ε, πιο παραδόξως η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου όλοι συμφωνούν ότι εμείς ερμηνεύουμε ορθά την συνθήκη της Λισαβόνας, ε, όχι το Συμβούλιο. Λοιπόν, ε, προς τα που κινείται η ισχύς όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι μέσα στις ομάδες εργασίας του Συμβούλιο μπορούν να επιτάσσουν και να αποφασίζουν ότι ε, σημεία κλειδιά αφαιρούνται από την πρόταση που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και να τα παραπέμπουν στο επόμενο Συμβούλιο αλλιώς Είναι σκανδαλώδες αυτό, είναι απαράδεκτο και ε, σε, αυτή την, ε, αυτό το διαθεσμικό αγώνα ε, ο Πάτε Γκάλεχερ ανέβαλε την τελική ψηφοφορία για τον κανονισμό τεχνικών μέτρων πετώντας το γάντι στην Επιτροπή και το Συμβούλιο για να ξεμπλέξουν αυτό το κουβάρι και πρέπει να σας πω ότι τώρα μας έχουν θέσει μπροστά σε ένα τελεσίγραφο ε, και η συγχύτρια καλά θα έκανε να ε, ολοκληρώσει παρόλα αυτά την ε, έκθεσή της και πρόεδρε πραγματικά πρέπει να εξετάσουμε άλλα εναλλακτικά μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να περάσουμε ένα σαφές και ηχηρό μήνυμα προς το Συμβούλιο ότι δεν δεχόμαστε τέτοιου είδους πάυση, διακοπή των δραστηριοτήτων του Κοινοβούλου. Ευχαριστούμε κύριο Βαλέσα παρακαλώ. E, Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Στην προηγούμενη συνεδρίαση συμφωνήσαμε όλοι ότι ο κανονισμός αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα σχεδίου διαχείρισης των αποθεμάτων μπακαλιάρου απολύτως μη ρεαλιστικό. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Ντότζ για την ενδελεχή προσέγγιση και ανάλυση του ζητήματος. Η αναθεώρηση του σχεδίου πρέπει να ακολουθεί τις νομικές ε, συμβουλές και αυτό είναι πολύ σημαντικό μου φαίνεται σαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθεί να απλουστεύσει τους κανόνες αλλά ουσιαστικά να τους καθιστά ακόμα πιο σύνθετους και το παράδειγμα που θα δώσω είναι το άρθρο 11α το οποίο δυστυχώς περιλαμβάνει πολλούς ασαφείς όρους και εκφράσεις συνεπώς θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η μία αφορά τα κριτήρια Υπάρχουν τρία κριτήρια που απονομάζονται εκεί και ε, υποτίθεται ότι πρέπει να συμμορφωνόμαστε, να συμμορφωνόμαστε με όλα αυτά ή με ένα από αυτά. Δεύτερον, πόσο καιρό θα ισχύει η εξαίρεση. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το πόσο υποτίθεται ότι θα παραμένει σε ισχύ και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται. Θα ήθελα να υποστηρίξω την κυρία Ντότς και να επικρινώ την ιδέα που επέκρινε και ο κύριος Στίβενσον μια ιδέα που έχει μόλις ανακύψει και που δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κανείς δεν μας έχει πει επίσημα για τη διαγραφή των άρθρων 9 και 12, το οποίο είναι απίστευτο. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να το ε, επισημάνουμε, όπω έκανε και η κυρία Ντότζ και συμφωνώ μαζί τη ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε το σχέδιο στο σύνολό του και να συμπεριλάβουμε τα άρθρα στην έκθεση, τα άρθρα τα οποία προσπαθεί να, να, εξαιρέσει το... να διαγράψει το Συμβούλιο. Αυτό που κάνει το Συμβούλιο δεν βοηθά στην αποφυγή της κρίσης. Αντιθέτως, καθιστά τις σχέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων ακόμη χειρότερες και θα πρέπει να το καταδικώσουμε όλοι και χαίρομαι που όλοι συμφωνούμε από αυτήν την άποψη. Ευχαριστώ. Η κυρία Φράγκα, ακούστε, δεν θα ασχοληθώ με την ε, ουσία του θέματος. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα, απο, τα αποτελέσματα για τον Βακαλό. Το σχέδιο ανάκτησης ε, του του ερυθρού τόνου είναι τόσο βρετικά που δεν θα ασχοληθώ. Από θεσμικής πλευράς. Μέχρι ποτέ εμείς θα συνεχίζουμε να ε, υπομένουμε αυτή την κατάσταση με την θέση του Συμβουλίου. Δική μας είναι η ευθύνη, διότι δεν είμαστε σε θέση να ακολουθήσουμε ένα θεσμικό σχέδιο σε σχέση με τους άλλους. Τι κάνουμε, καθυστερούμε τις ε, ψηφοφορία των εκθέσεων, το έχω πει 20 φορές τουλάχιστον. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να σταματήσουμε τη μεταρρύθμιση. Διότι το θέμα του βασικού κανονισμού στη μεταρρύθμιση βασίζεται σε χόρτιο δεσμό, κυρίως για τα σχέδια διαχείρισης. Και αν εκ των προτέρων δεν μπορέσουμε το θεσμικό πρόβλημα με το Συμβούλιο να το επιλύσουμε, και δεν συμφωνώ με τον κύριο Στίβενσον, όλοι οι υπουργοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι δημοσίες δεν θέλουν να το αναγνωρίσουν. Συνειδητοποιούν όμως όλοι οι δημοσίες που είναι το πρόβλημα. Αν λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αλληλείας δεν ασχοληθεί με το θέμα αυτό, ό,τι μας αξίζει θα έχουμε. Διότι θα ληφθούν και αποφάσεις που πάνε και πάρα πολύ πιο μακριά από το 43-3 σύμφωνα με την ε, σύνδεξη της Λισαβόνας. Το θέμα δεν είναι ε, θέμα... Το θέμα είναι μόνο θέμα συναρμοδιότητας στα πλαίσια του 43-2. Εγώ 20 φορές πρότεινα να σταματήσει αυτή η μεταρρύθμιση, διότι είναι ο μόνος τρόπος για τον οποίο και η Κομισιόν και το ε, Συμβούλιο θα ε, καταλήξουν σε συμφωνία μαζί μας. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει, εάν δεν λύσουμε το θεσμικό θέμα, επαναλαμβάνω, να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση. Όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι και οι συντονιστέ και όλοι. Ή λοιπόν θα πρέπει να πάρουμε τώρα απόφαση ή θα μα συμβεί ότι μα αξίζει. Και προφανώς το Συμβούλιο μας έχει γράψει στα παλιά του υποδήματα. Εάν λοιπόν εμείς δεν ενεργήσουμε με αποφασιστικότητα και σοβαρότητα για να μπλοκάρουμε το βασικό κανονισμό, δεν θα κάνουμε τίποτε. Θα συνεχίσει να κάνει ό,τι του γουστάρει το Συμβούλιο και επαναλαμβάνω θα πέσει επί της κεφαλής μας ό,τι μας αξίζει. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει καμία άλλη παρέμβαση. Ο κύριος Γκάλαχερ. Δεν θα μιλήσω πολύ. Ουσιαστικά θα επαναλάβω κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε κάποιο αδιέξοδο. Βάσει των πληροφοριών που ακούμε και όλοι το γνωρίζαμε ήδη, το Σύμβουλο προσπαθεί να το παρακάμψει αυτό βγάζοντας κάποιες πτυχές ώστε να μπορεί να ληφθεί κάποια απόφαση στην Επιτροπή αποφασίσαμε ουσιαστικά τι πρέπει να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να το υποδείξω εδώ σε μια δημόσια συνεδρίαση, αλλά πρέπει να αναλάβουμε δράση. Θεωρούμε δεδομένο και επαναλαμβάνομαι, το Συμβουλίο δεν αναγνωρίζει τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει εμείς να συμμορφώνομαστε δηλαδή με τους κανονισμούς της Λισαβόνας, αλλά αυτοί όχι είχαμε προβλήματα στις δικές μου εκθέσει και του κυρίου Στίβενσον και στα, μακροπρόθεσμα, στα σχέδια μακροπρόθεσμης διαχείρισης γιατί κάθε δύο εβδομάδε πρέπει να ερχόμαστε εδώ και να ε, προσπαθούμε τόσο πολύ να έχουμε βιώσιμη αλία. Πώς θα το κάνουμε αν δεν έχουμε σχέδια μακροπρόθεσμης ε, διαχείρισης. Θα πρέπει να ε, επιτείνουμε τις προσπάθειές μας και να δηλώσουμε ότι χάρη στις δράσεις που έγιναν την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν κάποια επικίνδυνα ζητήματα ελέγχου. Αυτό δεν ήταν δική μου απόφαση, ήταν ομόφωνη απόφαση άλλον και αν το Συμβούλιο δεν το αναγνωρίσει αυτό θα χρειαστεί να αναθεωρήσουμε και τη θέση μας και τη σχέση μας μαζί τους. Ευχαριστώ. No, I won't take a lot of time. Η κυρία Λέβιν, ναι, και εγώ σύντομη θα είμαι. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ντότζ ε, για την εργασία της. Ε, είμαι σκιώδης για τους πρασίνους και θα παρακολουθήσω από κοντά το θέμα. Ήθελα να τονίσω πάντως ότι υπάρχει πλήρης ομοφωνία ε, για την απόφαση αναβολής τελικής ψηφοφορίας του κανονισμού των τεχνικών μέτρων στην Ολομέλεια την εβδομάδα που μας πέρασε και ότι συμφωνούν όλα τα μέλη της Επιτροπής ότι πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα των μακροπρόθεσμων σχεδίων διαχείρισης και το θέμα των, της κατανομής των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ με την κυρία Φράγα ότι πρέπει να ε, δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το ζήτημα, κυρίως εν ώψη και της μεταρρύθμιση μεταρρύθμισης αλληλευτικής πολιτικής. Ε, δεν νομίζω ότι παρακρατώντας, ε, μάλλον έχοντας αυτή την παραγγελιστική συμπεριφορά για τα μακροπρόθεσμα σχέδια, λύνεται το πρόβλημα. Το Συμβούλιο πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να μας πάρει στα σοβαρά. Δεν μπορούμε απλώς να παρακολουθούμε σε εξελίξεις εκεί. Ευχαριστούμε κυρία Λοβίν. Ευχαριστώ. Άκουσα τι είπατε και πρέπει να πω ότι γενικά συμμερίζομαι όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν. Απλώς θα ήθελα να αποσυμφωνήσω το εξή. Πολλά λέμε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Αύριο θα θέσουμε το θέμα της συνάντηση των συντονιστών, διότι όντως τα τελευταία εννέα δεν είναι ε, θετικά. Αντιθέτως, είναι ανησυχητικά. Και στις 18 Δεκεμβρίου προβλέπει το Συμβούλιο να αλλάξει κάποια στοιχεία από την πρόταση αυτή όσον αφορά τα ε, και δεν μπορούμε να περιμένουμε και να έχουμε σκαμπανεβάσματα σε αυτό που θα κάνουμε. Δηλαδή, εμείς να είμαστε κομπάρσι, να αφήσουμε το Συμβούλιο να κάνει ό,τι θέλει μόνος του και να μας αγνοεί, να μην μας εμπιστεύεται και να αγνοεί και την ίδια τη συνθήκη και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι χάσαμε πολύ περισσότερο από ό,τι και με τα πολυετή σχέδια. Νομίζω ότι το συζητήσαμε αυτό διεξοδικότατα, αυτό το οποίο ζητώ κυρίως στου συντονιστέ, ε, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους που δεν είναι συντονιστέ, αλλά να το αναφέρουν στους δικού τους συντονιστές, αύριο να δουν τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Διότι όντω η απόφαση να μην ψηφίσουμε στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα. Καλό ήταν έως χειρονομία, αλλά δεν έγινε καμία κίνηση υπέρ της επίλυσης του όλου θέματος. Αντιθέτως, πρέπει να πω ότι έγιναν πιο ριζοσπαστικοί όσον αφορά τη θέση του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε κάποια απόφαση και την άποψή μου αναμφίβολα το καλύτερο θα είναι οι βουλευτέ σήμερα και αύριο οι συντονιστέ να μπορέσουμε να δούμε αν θα πάρουμε μία κάποια απόφαση ή να σταυράσουμε τα χέρια και να περιμένουμε. Διότι ό,τι κάναμε τώρα δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Αύριο λοιπόν, αύριο λοιπόν θα συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Θέλει να προσθέσει κάτι η Επιτροπή, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Κυρία Μονσένη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε την κυρία Ντόντ για την πολύ επικοδομητική έκθεση και ανάλυση της κατάστασης. Επιτρέψτε μου να κάνω μερικά σχόλια. Όσον αφορά την πρόταση της ε, Επιτροπής, έχει καθυστερήσει, αλλά την πραγματικότητα δεν καθυστερήσαμε. Ήταν μακροχρόνια η διαδικασία αξιολόγησης και ανάλυσης του γιατί αυτό το σχέδιο δεν λειτουργεί. Φυσικά υπάρχει πρόβλημα στην νομοθεσία, στον ίδιο, στους κανονισμούς και υπάρχουν και πολλά προβλήματα υλοποίηση αυτού του μακροπροθεσμού σχεδίου διαχείριση. Ήταν λοιπόν μακροσκέληση διαδικασία συζητήσεων για τα αποτέλεσμα των αξιολογήσεων με τα κράτη-μέλη, με τους ενδιαφερόμενους, με τη βιομηχανία για να ε, καταφέρουμε να βρούμε την καλύτερη λύση για το επόμενο βήμα όσον αφορά αυτό το σχέδιο. Πρόκειται για μια μακροχρόνια εργασία, ένα νέο σχέδιο διαχείρισης και ένα σχέδιο, νέο σχέδιο αλληλευτικό. Σήμερα καταλήγουμε στο τελικό αποτέλεσμα ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα πρόταση σχεδίου μεικτών, μεικτής αλίας. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι μετά από ένα νέο γύρο διαβουλεύσεων με τα κράτη-μέλη και του ενδιαφερόμενου να προτείνουμε αυτή την τροποποίηση η οποία προσπαθεί στα γρήγορα να διορθώσει κάποια, να επιλύσει κάποια προβλήματα βραχυπρόθεσμα. Αλλά τώρα έχουμε αυτή την τροπολογία. Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αυτή η πρόταση θα μπορούσε να τροποποιηθεί και ότι θα ήταν δυνατή η επιτευξή του απότερου στόχου που τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουν να επιτύχουν, δηλαδή το να παγώσουν τις προσωστώσεις για το επόμενο χρόνο ώστε να υιοθετηθεί γρήγορα αυτή η τροπολογία. Τώρα εγώ κατεγράψα τις αντιδράσεις σας λαμβάνοντας υπόψη και το τι συμβαίνει στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η συζήτηση στο Συμβούλιο βρίσκεται ακόμα σε επίπεδο ομάδας εργασίας. Το Συμβούλιο λοιπόν δεν έχει ακόμα καταλήξει σε επίσημη απόσταση, ε, απόφαση θέσης φυσικά. Ακούγονται φήμες ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να επιτευχθεί ομοφωνία, αλλά η Κομισιόν εξακολουθεί να πιστεύει ότι ίσως αυτό να μην αληθεύει. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι η εμπλοκή στα θεσμικά όργανα και οι συνέπειες αυτής της πιθανής θέσης του Συμβουλίου δημιουργούν ένα σημαντικό θεσμικό πρόβλημα και διένεξη μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Πρόκειται για κάτι που γνωρίζουν οι πρωτεύουσες. Δεν είμαι βέβαιη λοιπόν η Κομισιόν, δεν είναι βέβαιη ότι θα επιτευχθεί ομοφωνία. Γνωρίζουμε ότι γίνονται πολλές συζητήσεις μεταξύ ομάδων εργασίας ομάδες εργασίας και πρωτευουσών. Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε, να ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει ομοφωνία και θα αναλάβει το Συμβούλιο μια πιο υπεύθυνη προσέγγιση. Πιστεύω ότι πρέπει να παραμένουμε ανοιχτό μυαλί και να δούμε ποια θα είναι η τελική θέση του Συμβουλίου. Φυσικά η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφής. Θεωρούμε ότι η πρόταση της Προεδρίας στο Συμβούλιο για τη διχοτόμηση της πρότασης δεν βρίσκει νομική βάση στη συνθήκη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του σημερινού σχεδίου θα πρέπει να ε, να τεθεί στο πλαίσιο της ε, συνήθους νομοθετικής διαδικασίας όπως ορίζεται από το σχετικό άρθρο στη συνθήκη. Φυσικά οποιαδήποτε θέση που ενδεχομένως θα λάβει το Συμβούλιο όσον αφορά τη διχοτόμηση της πρότασης θα εξεταστεί, θα θεωρηθεί παράνομη από την Κομισιόν. Αλλά επαναλαμβάνω ξανά, δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα λάβει θέση. Στο τρέχον λοιπόν ε, περιβάλλον εμείς είμαστε ανοιχτοί προς το Κοινοβούλιο και δείχνουμε στο Συμβούλιο ότι πρέπει να προχωρήσει και να ασκήσει τα καθήκοντά του. Ε, η Επιτροπή αυτή μπορεί να προχωρήσει και να εκφράσει την υποστήριξή της ε, για την πρόταση της Κομισιόν. Σε αυτή την περίπτωση για να μην χάνουμε από τα μάτια μας τον απότερο σκοπό της πρότασης, εάν το Συμβούλιο δεν καταλήξει ομοφωνία, και εμείς αυτό ελπίζουμε, και επανέλθει στην πρόταση της Κομισιόν, εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα αυξημένη ευελιξίας των προσπαθειών για τα συνολικά επιτρεπόμενα λιεύματα. Πιστεύω λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι έτοιμο να αντιδράσει σε αυτή την πρόταση με τρόπο τέτοιο, ώστε σε περίπτωση μη επίτευξη ομοφωνία στο Συμβούλιο η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου να είναι έτοιμη και το Κοινοβούλιο να δείξει, να αποδείξει την ικανότητά του να υλοποιήσει τα καθήκοντά του, ότι θα έχει μια πρόταση έτοιμη για έγκριση στις αρχές του επόμενου έτους. Εάν η πρόταση μπορέσει να υιοθετηθεί αρχές του επόμενου έτους, τότε θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τον απότερο στόχο της παρούσας πρότασης, δηλαδή να εφαρμόσουμε αναδρομικά το πάγωμα της αλληλευτικής προσπάθειας από την 1η Ιανουαρίου του 2013. Εξακολουθούμε λοιπόν να πιστεύουμε ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση και εμείς υποστηρίζουμε τόσο το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε σίγουροι ότι και τα δύο θεσμικά όργανα θα εξακολουθήσουν να αναλύουν και να λαμβάνουν αποφάσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της απόφασης της Κομισιόν εξασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή υιοθέτηση της πρότασης αυτής. Εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες για συγκεκριμένα άρθρα του κανονισμού. Θα ζητήσω λοιπόν από τους συναδέλφους μου να μπουν σε περισσότερες λεπτομέρειε να σχολιάσουν τα συγκεκριμένα άρθρα αυτά. Θα ήθελα πρώτα να αντιδράσω στα σχόλια για το ζήτημα των απορρίψεων των απορριπτόμενων αλλιευμάτων να υπογραμμίσω ότι σε αυτή την πρόταση δεν περιλαμβάνεται απαγόρευση απορριπτόμενων ελευμάτων για τον μπακαλιάρο. Απλά υπάρχει μια υπενθύμηση στο άρθρο ότι τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των απορριπτόμενων αλλιευμάτων, διότι τα απορριπτόμενα αλλιεύματα μπακαλιάρου βρίσκονται ακόμα σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο και αν δεν καταφέρουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα των απορρίψεων δεν θα καταφέρουμε ποτέ να λύσουμε το πρόβλημα της θνησιμότητας των αυτού του αποθέματος. Όποιοι λοιπόν και αν είναι οι κανόνες αυτού του σχεδίου, αν δεν καταφέρουμε να μειώσουμε το επίπεδο απορρίψεων, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να μειώσουμε τη θνησιμότητα των αποθεμάτων αυτών. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω τώρα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις για το άρθρο 11 μακρά η ιστορία της εφαρμογής του άρθρου 11 υπάρχει η αρνητική αντίληψη ότι δεν γίνεται να αποκλείσουμε από το καθεστώς αλλιευτικών προσπαθειών κάποια σκάφη. Ε, ως προς τη συλλογή δεδομένων επιστημονικών στοιχείων, σκάφη που κάνουν ε, τις δοκιμές, ε, in year and also ε, παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα, ε, ε, δεν είναι όμως ουσιαστικές οι επιπτώσεις και γι' αυτό αποφασίσαμε να απλουστεύσουμε το άρθρο και νομίζω ότι η τωρινή του μορφή είναι απλοποιημένη. Όπως μας υπέδειξαν οι επιστήμονες, ο ο αποκλεισμός του άρθρου 11 μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε περιπτώσεις όπου είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το απόθεμα γάδου. Δεν μπορούμε όμως να προκαθορίσουμε ποιες είναι αυτές οι περιοχές. Χρειαζόμαστε πιο ευέλικτη προσπάθεια, δηλαδή η Οικονομική, Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή θα εξετάζει κατά περιοχή και θα δίνει τις συμβουλές του. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο παλιό και το νέο προτινόμενο σύστημα ε, και μπορούν ε, νέα σκάφη και νέα κράτη-μέλη να ζητήσουν χορήγηση αυτού του ειδικού καθεστώτος. Ε, προς το παρόν ε, ασχολούμαστε με συγκεκριμένα κράτη-μέλη και συγκεκριμένες ομάδες σκαφών. Τώρα με τη νέα πρόταση ο αποκλεισμό η εξαίρεση θα διευρυνθεί για να καλύπτει παραδείγματο χάρη επιλεκτικό αλλιευτικό εξοπλισμό και οποιοδήποτε κράτος και σκάφος χρησιμοποιήσει αυτόν τον επιλεκτικό μηχανισμό μηχανισμό ε, θα δικαιούται την εξαίρεση. Θα είναι μια γενική εξαίρεση. Δεν υπάρχει ω εκ τούτου χρονοδιάγραμμα. Δεν αποκλείουμε συγκεκριμένα σκάφη, αποκλείουμε περιοχές και συγκεκριμένο αλλιευτικό εξοπλισμό και επιστημονικό ώστε πυριώνεται ότι κάτω από τα 300 μέτρα ε, βάθους εννοούμε δεν υπάρχουν ε, αποθέματα γάδου, δεν, είναι δυνατός ε, ο αποκλεισμό, η εξαίρεση και χρειάζεται έλεγχο και γι' αυτό κάνουμε την πρόταση αυτή μέσα στο άρθρο 11. Μπορούμε όμω να μπούμε και σε λεπτομερέστερε διευκρινήσει. Αν κάποιο βουλευτή επιθυμεί να κατανοήσει καλύτερα την λειτουργία αυτού του μηχανισμού. Μπορούμε με περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες να διευκρινίσουμε τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού, εάν το επιθυμείτε. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ποιο ζητάει το λόγο, η κυρία Ντότς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Περίμενα με ανυπομονησία να ακούσω και τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, αλλά δεν εκπροσωπείται το Συμβούλιο εδώ στην αίθουσα για την εξέταση του σημείου. Λοιπόν, θα επαναλάβω αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση και η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ακριβώς τι σκοπεύει να κάνει. Κατά τη δική μου άποψη πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει η έκθεση όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά γρήγορα και πρέπει να αποδείξουμε εμπράκτος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να λάβει υπόψη τις επιστημονικές συμβουλές, να ακούει την άποψη της βιομηχανίας και να εξασφαλίσει έτσι μεγαλύτερη ευελιξία. Χρειαζόμαστε δε λεπτομερέστερες ε, ε, ε, διατάξεις και όχι μόνο μια απλή απαλήφη του άρθρου 9 και 11 για να μπορέσουμε τελικά να εγκρίνουμε τον κανονισμό. θα ε, εξετάσει η Επιτροπή μας αν μπορούμε να επισπεύσουμε την έγκριση της έκθεσης. Ε, πάντως ε, είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να καταθέσετε νέες θέσεις με ιδέες ε, για να βελτιώσουμε την έκθεση. Μπορείτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία να έρθετε σε επαφή ε, μαζί μου. Θα δούμε σε κάθε περίπτωση και ποια θα είναι η έκβαση της ψηφοφορίας στην Κορεπέρ και θα δράσουμε αναλόγως στην συνέχεια. Ευχαριστούμε ο Αντιπρόεδρος ε, Στίβενσον. Ένα σύντομο σχόλιο, ακούγοντα όλα αυτά που λέει η Κομισιόν, ότι πολύ λόμπινγκ λαμβάνει η χώρα στις πρωτεύουσε των χωρών ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία για αυτό το ζήτημα στο Συμβούλιο. Αναρωτιέμαι, επειδή εδώ ουσιαστικά συζητάμε μεταξύ Κομισιόν και Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο παραμένει λίγο άμετοχο Αναρωτιέμαι κατά πόσο οι συντονιστέ αύριο θα μπορούσαν να εξεταστούν το ενδεχόμενο συγγραφή μια επιστολή από εσά, κύριε Πρόεδρε, προ όλου του Υπουργού Αλία, ε, στην οποία θα εκφράζονται οι ανησυχίε μα για το ζήτημα και ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε με ρεαλιστική μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική, εάν συνεχίζουν να μα μπλοκάρουν σε αυτά τα ζητήματα αυτέ οι ε, διενέξει μεταξύ θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ κύριε Στίβεν. Σας ευχαριστώ για την καλή σας φούτσα, αλλά 27 επιστολές σε αυτούς που έχουν πολύ σαφείς ιδέες για το τι μπορούν να κάνουν, δεν θα έχει και μεγάλο όφελος. Τώρα, όπως είπαμε, εδώ και πολύ καιρό υπάρχουν κάποια ε, σχέδια για τα οποία δεν έχουμε λάβει αποφάσεις. Έχουν παραλύσει τα πάντα κοινοβούλια. Δεν υπάρχουν αποφάσεις διότι ε, κάποιες ε, αποφάσεις ε, όταν ληφθούν θα μας οδηγήσουν σε προσφυγή στο δικαστήριο μας. Εν πάση περιπτώσει την πρότασή σας ε, θα την μεταφέρω αύριο, αλλά δεν νομίζω ότι παρά την καλή της θεωρητική αξία θα έχει μεγάλα πρακτικά αποτελέσματα. Τώρα, θα ήθελα να περάσω στο σημείο 8, αλλά πριν θα ήθελα να χαιρετήσω τους εκπροσώπους της Γαλλικής Σχολής Ασφάλειας στη Θάλασσα της Γαλλίας. Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Σημείο 8. Απόφαση Επιτροπή Δικοινοποίηση Τρίτων Χωρών που η Επιτροπή θεωρεί πιθανό να χαρακτηριστούν ω μη συνεργαζόμενε τρίτε χώρε δυνάμει του κανονισμού 1005 περί δημιουργία κοινοτικού συστήματο πρόληψη αποτροπή και εξάλληψη παράνομη λαθρέα και άναρχη αλήθεια. Όπω ξέρετε, αυτό ο κανονισμό θέλει να εντοπίσει τις χώρες αυτές. Το θέμα αυτό συζητήθηκε και πρόσφατα. Η συγγετής είναι ο κύριος Ρωμέβα και η Επιτροπή σε αυτή την περίπτωση με δική της πρωτοβουλία μας ζήτησε να συμμετάσχουμε σε αυτή την συνεδρίαση. Εμείς με την καλύτερη δυνατή διάθεση το κάναμε για να δούμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε αυτές τις τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στις ε, ε, νόμιμες διαδικασίες Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πέρνης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, είπατε, την προηγούμενη 15 Νοεμβρίου ενέκρινε μία απόφαση η Επιτροπή με την οποία κοινοποιείται σε 8 χώρες η δυνατότητα να θεωρηθούν ως χώρες που δεν συνεργάζονται στο πνεύμα της ε, εξάλληψης της παράνομης και αρχές αλία. Φίτζι, Καμπότζη, Γκινέα, Παναμά, Σρι Λάνκα, Τονγκό και Βανουάτου λόγος για τον οποίο η Επιτροπή αποφάσισε καταρχάς να, ε, να απευθυνθεί σε αυτές τις τρίτες χώρες που δεν συνεργάζονται είναι διότι έχει αποδείξεις και δεν επομίζονται τις ευθύνες τους ως χώρες εμπορίας, χώρες σημείας, χώρες παράκλησης. Άρα δεν επομίζονται, όπως είπαμε, με κατάλληλο τρόπο τις ευθύνες τους και δεν τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή έκανε μία πάρα πολύ εμπεριστατωμένη και εκτεταμένη ανάλυση που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια με στόχο αφενός να μπορέσει όλες τις αποδείξεις και τις μαρτυρίες να τις συλλέξει ώστε από νομικής απόψεως και πολιτικής απόψεως να έχει βάσιμα στοιχεία και δεύτερον για να δώσει χώρες αυτές τη δυνατότητα να αρχίσουν να ασκούν σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης τα ε, δικαιώματά τους και να σέβονται τους κανόνες με ικανοποιητικό τρόπο. Ο κατάλογος των χωρών που έχετε εδώ, αυτές οι 8 χώρες, πρέπει να πω ότι δεν είναι όλες οι χώρες τις οποίες, ε, ε, για τις οποίες έκανε έρευνα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών η Επιτροπή. Πράγμα το οποίο υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όταν κάνουμε κρίσεις και αξιολόγηση αυτών των οποίων κάνει στα πλαίσια της παράνομης αλληλείας ή ε, δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο ποιες χώρε είναι σε αυτόν τον κατάλογο, αλλά και ποιες δεν είναι και για ποιο λόγο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι η απόφαση που η Επιτροπή τώρα μόλις υιοθέτησε δεν σημαίνει ότι θα υπάρξουν εμπορικές κυρώσεις. Πρόκειται για προεντοπισμό αυτών των χωρών και αμέσως μετά ποια είναι η επίπτωση καλείται η εν λόγω χώρα να αρχίσει ένα σχέδιο δράσης για να αλλάξει τις αδυναμίες και τα προβλήματα που έχει όσον αφορά τον έλεγχο του ελευτικού της στόλου και της δίδεται σε έξι μήνες η δυνατότητα της χώρας αυτής να επιλύσει τα προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν με σαφήνεια. Δεν πρόκειται λοιπόν για κύρωση, αλλά για προειδοποίηση που έχει σημαντική πολιτική και νομική ε, χρειά για να μπορέσουμε στην ευρωπαϊκή κοινότητα να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλληλεία. Εάν δεν μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή από τις χώρες αυτές το σχέδιο δράσης, και εφόσον έχει δοθεί αυτό το μήνυμα το νομικό και το πολιτικό, κινδυνεύουν να υποστούν και εμπορικές κυρώσεις οι χώρες αυτές, διότι όπως ξέρετε στα πλαίσια αυτού του κανονισμού υπάρχουν απαγορεύσεις εισαγωγών προϊόντων αλίας παράνομης, ε, καταγγελίας των αλληλευτικών συμφωνιών ή απαγόρευση ε, με αυτών, σκαφών με σημαία αυτών των χωρών που μπορούν να αλλιεύουν αλλού. Όλα αυτά έχουν γίνει με πάρα πολύ εμπεριστατωμένους ελέγχους εκ μέρους της Επιτροπής για να δούμε αν μπορούν τέτοιου είδους σχέδια να τεθούν σε εφαρμογή. Και μετά από 6 μήνες θα είμαστε σε θέση να κάνουμε εκτίμηση του γεγονότος Ε, εφαρμογής αυτών των μέτρων που προτείνουμε πριν να αρχίσουμε σε αρνητική περίπτωση να εφαρμόσουμε εμπορικές κυρώσεις. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν και πολλές περισσότερες χώρες στη δουλειά της Κομισιόν από αυτές τις οκτώ που αναφέρονται εδώ. Κατά έργα των δύο τελευταίων ετών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε στις έρευνες που κάνει να κάνει η ιεράρχηση των ε, προτεραιοτήτων κυρίως για τις χώρες τις οποίες υπάρχουν πολλές σημαίες ευκαιρίες. Υπάρχουν πολλά στοιχεία όσον αφορά τον κανονισμό αυτό με την παράνομη αλληλεία, αλλά αυτό κυρίως που μας απασχόλησε, όπως σας είπα, είναι να μπορούμε να δούμε τι γίνεται στις χώρες που δίνουν ε, σημαίες ευκαιρίες, που πολλές φορές δεν έχουν εμπορική αγορά, δεν έχουν τεχνογνωσία, δεν έχουν παράδοση στην αλληλεία και παρόλα αυτά έχουν στα μητρώα τους ένα δυσανάλογο αριθμό ε, σκαφών στο οποίο έχουν χορηγήσει σημαίες ευκαιρίε χωρίς να μπορούν να διαχειριστούν το όλο σύστημα. Αν αυτές οι χώρε οι οκτώ έχουν κάτι το κοινό είναι το ότι έχουν στα μητρώα τους πάρα πολλά αλλιευτικά σκάφη τα οποία δεν μπορούν όντω να ελέγξουν ή να ασκήσουν αποτελεσματικό κανέναν έλεγχο για να μπορέσουν να τηρήσουν τους κανόνες που ισχύουν μετά την χορήγηση της σημαίας που χορήγησαν. Θα ήθελα να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Στην Ινδονησία, Φερρυπίν, όλες οι, ε, ό,τι έκανε, όλες οι δράσεις ε, που ανέλαβε η Κομισιόν έδωσαν από την τρίτη χώρα αυτή ε, πάρα πολλά ε, θετικά αποτελέσματα, δράσεις και μέτρα για να αλλάξει η κατάσταση και όταν είδε η Κομισιό ότι μια χώρα που αποτέλεσε αντικείμενο ερευνών τα δύο τελευταία χρόνια αντέδρασε θετικά, αποφάσισε να μην το συμπεριλάβει στον κατάλογο. Γιατί, διότι τελικά ο ίστατος στόχος αυτού του κανονισμού δεν είναι να επιβάλλουμε κυρώσεις στις χώρες, αλλά δεν είναι να απαγορεύσουμε τις εισαγωγές. Ο ίστατος στόχος είναι να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά κάποιων χωρών ώστε να συμπεριφέρονται σοβαρά και όταν χορηγούν την σημαία σε κάποια σκάφη να μπορούν να το κάνουν τηρώντας τους κανόνες του ε, δικαίου της θαλάσσης. Και αυτό που είναι ευχάριστο είναι να μπορούμε από τον κατάλογο αυτό να αφαιρούμε χώρες που συμπεριφέρονται σωστά. Αναμφίβολα κύριε Πρόεδρε, θα διαρωτηθείτε τώρα τι γίνεται. Σε σχέση με τις χώρες αυτές όπως σας είπα, υπάρχουν δύο μεγάλες ε, ε, γραμμές δράσης. Για αυτά τα οχτώ κράτη που εντοπίσαμε καταρχάς, η Κομισιό πρότεινε σχέδιο δράσης και η εργασία των υπηρεσιών της Επιτροπής του επόμενους 6 μήνες θα συνίσταται στο να παρακολουθούμε τι γίνεται και να αρχίσουμε διάλογο με τις εν λόγω χώρες για να δούμε αν όντω πράγματι είναι σε θέση και έχουν την πολιτική βούληση και διαθέτουν τα μέσα για να μπορέσει αυτό το σχέδιο δράση να εφαρμοστεί. Αυτή θα είναι η μεγάλη προτεραιότητα του επόμενου εξάμεινου. Αλλά θα πρέπει επίση να προσθέσω ότι η δράση τη Επιτροπή δεν σταματά εδώ. Θα, μου ερωτήσετε, θα με ρωτήσετε το εξή. Όλε δυνητικά οι χώρε μπορούσαν να κάνουν παράνομη εργασία, όχι απαραίτητο. Άρα, παραλίλου η Επιτροπή θα συνεχίσει κατά τη διάρκεια όλου του επομένου έτους τις ε, συμπεριρωματικές έρευνες. Υπάρχει μια σειρά χωρών, τρεις υπήρους στην Ασία, στην Αφρική και στην Αμερική που θα ερευνήσουμε για να δούμε ενδεχομένως μήπως θα, μπορούσαμε, να καταρτήσουμε ένα δεύτερο κατάλογο του 2013. Δεν ε, είναι πολύ αρχή ακόμη, δεν μπορώ να σας πω ποιες θα είναι οι χώρες αυτές. Το υπάρχει ε, αυτή τη στιγμή προσπάθεια να ολοκληρώσουμε τα προγράμματα παρακολούθησης ε, των τυχών ανομαλιών στις χώρες αυτές και εκ με τα σχέδια δράσης για αυτές τις 8 χώρες θα συνεχίσουμε να ερευνούμε από την Κομισιόν και άλλες χώρες του κόσμου για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αν όντω υπάρχουν ε, βασικές ε, υπόνοιες και στοιχεία που θα μας οδηγήσει να συμπεριλάβουμε και άλλες χώρες σε λίστες. Θα σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο όπως ξέρουμε πάρα πολύ ενδιαφέρει την Επιτροπή σας και φαντάζομαι θα υπάρχουν και πολλές ερωτήσεις εν μέρους των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πένιες. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρωμέβα που είναι εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι τον κύριο Πένιες για την παρουσία του, αλλά διότι όπως κάναμε και σε προηγούμενες φορές, θα ήθελα να συγχαρώ την Κομισιόν για αυτό το βήμα προς τα πρός. Το περιμέναμε εδώ και πολύ χρόνο. Όντως, πρέπει να πω ότι στο ε, βήματα που έλαβε η Κομισιόν ανοίγουν ένα παραθυράκι για να ενεργήσουμε στον τομέα αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, συνειδητοποιούμε ούτως ή άλλως ότι εδώ έχουμε να κάνουμε, όπως είπε και ο κύριος Πένας, όχι με ένα κατάλογο για ακυρώσει, απλώς σηκώσαμε την κίτρινη κάρτα σε κάποιες χώρες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας κάνει να επιστήσουμε την προσοχή μας. Δηλαδή, δίνουμε κάποια μηνύματα σε κάποιες χώρες, καλό είναι αυτό, τους λέμε ότι θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά το θέμα αυτό, αλλά το θέμα ουσίας είναι να, να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα που θα εμποδίσουν συγκεκριμένα τέτοιου είδους πρακτικές. Χαιρετίζω λοιπόν αυτό το βήμα της Κομισιό και βεβαίως από αυτά που είπε η Κομισιό συμπεραίνω ότι αυτό είναι απόλυτα σαφές για αυτούς. Πρόκειται όμως για ένα σημείο εκκίνηση και δεν μπορεί να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Επιμένω λοιπόν ότι όλα αυτά που κάνουμε πρέπει να συνεχίζουν και με άλλα μέτρα. Έχουμε σε αυτό τον κατάλογο 8 χώρες που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ε, βεβαίως ε, μικρές χώρες. Σημαντικές ίσω, αλλά δεν έχουμε τα fish, τα μεγάλα ψάρια, του πιο σημαντικού. Δεν έχουμε εδώ τα ονόματα χωρών που είναι τόσο μεγάλες και σημαντικές και των οποίων οι επιπτώσεις τέτοιου είδους παράνομης αλληλείας είναι μεγάλες. Μελετώνται όλες αυτές οι χώρες, αλλά καλό θα είναι να ότι υπάρχουν χώρες την Ταϊβάν, την Κίνα, την Κορέα, την Ρωσία, τη Ρωσία με συγχωρείτε, που νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε όλους ιδιαίτερος. Όχι μόνον ε, η Κομισιόν, αλλά και το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τα προσέξουν ιδιαίτερα και να μην ε, λησμονούμε ότι η αξιοπιστία του καταλόγου αυτού επίσης εξαρτάται από το ποιες χώρες συμπεριλαμβάνονται και πρέπει να συμπεριληφθούν ε, όλες όσε ενέχονται σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλε χώρε. και ε, όπως είπε ο κύριος Πένι και εγώ κάνω αυτή τη θετική παρατήρηση. Θα, ε, πρέπει να υπάγονται σε έρευνα και πολλές άλλες ε, χώρες. Ε, λέμε λοιπόν και εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακαλούμε να διευρυνθεί ο κατάλογος και να συμπεριλάβει τις χώρες που και εγώ ανέφερα και άλλες που δεν ανέφερα. Ώστε όλοι τελικά να υπακούν στους ίδιους κανόνες. Κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό είναι το εξή. Τελικά θα είναι αξιόπιστος ο κατάλογος αυτός στο μέτρο που θα εφαρμοστούν κυρώσει. Και αυτό είναι κάτι Αξιοπιστή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει λοιπόν κάτι μόνο ω απειλή να το αναφέρουμε, θα πρέπει και να το εφαρμόσουμε. Θα πρέπει να είμαστε σαφεί. και αν θέλουμε να μπορέσουμε και εμεί με υποδειγματικό τρόπο να υπομισθούμε τι ευθύνε μα. Κατά κάποιο τρόπο θα δώσουμε να καταλάβουν και σε άλλες χώρες ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουν τέτοιου είδους πρακτικές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε συλλογικά με τις ε, ε συμβάσεις, με τις διεθνείς συνήθειες οι οποίες έχουν άμεση έμεση σχέση με το θέμα αυτό. Καθώς και με τις συμφωνίες που έχουν ε, ε, υπογράψει με χώρες περιοχής τους. Αναφέρομαι στον Παναμά, για να δώσω ένα παράδειγμα. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, θα πρέπει τέτοιου είδους ε, ε, ευθύνες που πρέπει να τις επομιστούν χώρες όπως ο Παναμάς, να τις αναφέρουμε. Και νομίζω ότι όσο μεγάλες κυρώσεις εμπορικές και να επιβάλλουμε, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας μπροστά σε κάποια θέματα τα οποία είναι οφθαλμοφανέστατα. Και μιλώ για τη Ρωσία και για την Κίνα. Εάν δεν πούμε με σαφήνεια περί τίνος πρόκειται και δεν εξηγήσουμε για ποιο λόγο μας ανησυχούν κάποιες πρακτικές, εάν δεν καταγγείλουμε ε, συγκεκριμένα ως Ευρωπαϊκή Ένωση τους μεγάλους ε, υπεύθυνου αυτών των πρακτικών, των αρνητικών που αντιμετωπίζουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Και όπως Είπα στην αρχή, θέλω να συγχαρώ και πάλι την Κομισιόν. Πρόκειται για ένα απαραίτητο και σημαντικό βήμα προ τα μπρο. Επιβεβαιώνω, όπω και η Επιτροπή, ότι είναι όμω ανεπαρκέ και ελπίζω ούτω ή άλλω ότι στον κατάλογο των χωρών αυτών θα μπορέσουν να προσθεθούν και άλλε κατάλογοι των σκαφών των αλληλευτικών για να ξέρουμε ποιοι είναι και οι κύριοι υπεύθυνοι. Διότι φοβούμε ή μάλλον. Έχω την ιδέα ότι... ότι μόνον έτσι θα έχουμε και μία πολύ πιο σαφή εικόνα για τις χώρες οι οποίες ε, προστρέχουν και προστατεύουν τέτοιου είδου πρακτικέ. Ευχαριστώ κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Κομισιό. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξη τον κύριο Ρωμέβα, διότι πιστεύω ότι η Κομισιό μέχρι τώρα είχε μία αμφίσιμη θέση. Απ' τη μια, μας δίνει κατάλογο χωρών που δεν συνεργάζονται και μετά επανέρχεται σε προηγούμενες αποφάσεις και δράσεις. Η συνεδρίαση έγινε στις 22 Οκτωβρίου στα πλαίσια της επιτροπολογίας και εκεί ξέρει ο κύριος Ρόμεβα ότι εκεί παίρνονται οι αποφάσεις με πλειοψηφία η Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλησε τον Μπελίζε να συμπεριληφθεί. Αυτό το θέμα με τις λίστες τι σημαίνει, ότι εμφαρμόζονται κάποια άρθρα ε, κυρίως όσον αφορά την εισαγωγή των ε, εισαγωγών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αυτό όμως συνειδητοποίησε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Πράγμα το οποίο δείχνει πόσο αμφίσιμες είναι κάποιες πολιτικές αποφάσεις. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανήλθε στις αποφάσεις της πολιτικής απόψεως και αυτό πρέπει να πω ότι είναι ούτως ή άλλως παράνομο και μίλησε για το άρθρο 31 που είναι η εντοπισμός ε, μη συνεργαζομένων χωρών. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε γίνει εκ των προτέρων, διότι όλοι ξέρουμε και συζητήσαμε πολλοί από εμά με τον Παναμά και ξέρουμε ότι ο Παναμάς ήδη είχε παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης κτλ. κτλ. Άρα το πρόβλημα είναι ότι η Κομισιό οπισθοχώρησε, διότι δεν ήθελε να εφαρμόσει το άρθρο 18 που είναι απαγόρευση εισαγωγών. Και εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Δεν την ενδιαφέρει αυτό το κανονισμό την Κομισιόν να την εφαρμόσει. Όχι μόνο γιατί δεν συμπεριλαμβάνει τις μεγάλες χώρες, αλλά δεν θέλει να εφαρμόσει και τίποτα εναντίον των μικρών χωρών. Εδώ και πολύ χρόνο ασχολούμαστε με αυτό το, χώρο, το θέμα. Και αν δεν εφαρμόζουμε το σχετικό κανονισμό, τι κάνουμε. Έκανε λοιπόν κάτι το παράνομο η Κομισιόν. Δεν ξέρω πώ να το πω, σω υπερβάλλω λέγοντα ότι έκανε κάτι παράνομο. Αλλά ε, οπισθοχώρησε τι αποφάσει που είχε λάβει πριν. Διότι έπρεπε στον κατάλογο αυτό να συμπεριλάβει και κάποια θέματα αποφάσεων του 2012 και αυτό θα είχε κάποιες επιπτώσεις και δεν θέλησε να το κάνει η Κομίσιο. Τώρα, το άρθρο 81 κατά την άποψή μου δεν ξέρω πόσο σημαντικό ήταν, διότι και στο παρελθόν Χίλιε φορές είχαν ζητήσει από αυτέ τις χώρες να παρουσιάζει το σχέδιο δράση τη. Δεν συμφωνώ με αυτό που έκανε η Κομισιόν. Νομίζω ότι πρόκειται για ε, πάρα πολύ σοβαρό παράπτωμα εκ μέρου τη. Και πάλι ο κανονισμός για την παράνομη αλληλεία δεν έχει καμία αξία. Παραμένει θεωρητικό στα χαρτιά. Και νομίζω ότι δεν είναι politically well τέτοιου είδους πράγματα να γίνονται. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την παρουσίαση. Ε, συμφωνώ με τα σχόλια των συναδέλφων και συγκεκριμένα τον κύριο Ρωμέδα ότι πρέπει να παραμείνουμε δική να διατηρήσουμε μια θετική αντιμετώπιση. Όμως, όπως σωστά είπε και η κυρία Φράγα, φαίνεται ότι κάποια κράτη-μέλη δεν επιδεικνύουν πολιτική βούληση. Αναφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον Μπελή. Ε, και είναι απαράδεκτο διότι έχουμε μια κυβέρνηση που λειτουργεί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προσπαθεί να προστατεύσει μια γνωστή σε όλους ε, σημαία βιτρίνα. Ε, ο κατάλογος αυτός σε κάθε περίπτωση είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα για την καταπολέμηση της ε, παράνομης άναρχης και λαθρέας αλίας και των αλλιευμάτων που εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για να ταυτοποιήσουμε, ας το πω έτσι, οικονομικούς φορείς της Ένωσης ε, που δραστηριοποιούνται με τέτοιες σημαίες. Η κυρία Φράγα αναφέρθηκε στον Πελίσε και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ ε, στην Σουηδία. Υπάρχουν τρεις εταιρείες ε, που έχουν την ε, ίδια σημαία Μπελής θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε κυρώσεις και να δηλώσουμε ότι δεν δεχόμαστε να εισέρχονται αυτά τα παράνομα λιεύματα στην Ένωση. Αυτό θα ήταν ένα ε, ε μείζον βήμα προς τα μπροστά και θα μια απτή απόδειξη ότι λειτουργεί ω ο κανονισμός. Ε, ο στόχος δεν είναι να επιβάλλουμε κυρώσεις σε τρίτες χώρες, είναι να ασκήσουμε πιέσεις σε οικονομικούς φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρησιμοποιούν τη σημαία αυτών των χωρών ούτως ώστε να συμμορφωθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει την πρωτοβουλία σύναψη ειδικών συμφωνιών με τη ΣΥΠΑ και την Ιαπωνία για να επιτύχει ένα συντονισμό αυτών των προσπαθειών. Έχουμε τις τρι, τους τρεις βασικούς αλλιευτικούς στόλους στον κόσμο κατά αυτόν τον τρόπο. Αν υπάρξει ε, συντονισμός ανάμεσα σε αυτούς τους αλλιευτικούς στόλους, τότε θα υποχρεώσουμε τους ε, ανεύθυνους ε, οικονομικούς φορείς ε, μέχρι σότου να εκλείψουν ε, οι σημαίες ε, βιτρίνα εν τέλει ε, πραγματικά κατά αυτόν τον τρόπο θα πιέσουμε τις εξελίξεις προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση. Σας συγχαίρω για τη δουλειά που έχετε κάνει, αλλά όπως σωστά είπε και η κυρία Φράγα, μπορείτε να βελτιώσετε ακόμη τα μέτρα που έχετε αποφασίσει. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι κάνει κάθε ό,τι περνάει από το χέρι της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, για τα σχέδια διαχείρισης. Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το βασικότερο πρόβλημα όταν εξετάσετε την περίπτωση αυτών των 8 χωρών. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα μπορούσαν να διορθώσουν. Ε, έχετε ελπίδες ότι τους επόμενους 6 μήνες ε, μπορούν να διορθώσουν κάτι. Αν δεχτούμε ένα σχέδιο δράσης, μήπως δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ποια είναι τα κριτήρια που θα ε, επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτω ώστε να διαγράψει αυτές τις χώρες από τον κατάλογο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Γκάλαχερ, παρακαλώ. Πρόεδρε, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Ε, τώρα που έχουμε την δυνατότητα συζήτηση ε, του πρωτοκόλλου ανάμεσα στην Μαυριτανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ω εκπρόσωπο τη Ιρλανδία δεν έχω κανένα συμφέρον ε, συγκεκριμένο για αυτέ τι διεθνεί συμφωνίε. Όμω, όπω είπε και η συνάδελφό, υποστηρίζουμε την βιωσιμότητα. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα ότι ίσως οι, οι διεθνείς συμφωνίες να διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη βιωσιμότητα της ε, ευρωπαϊκής αλλιευτικής πολιτικής, διότι πολλά σκάφη που αλλιεύουν σε διεθνή ύδατα που διέπονται από τα πρωτόκολλα αυτά, εάν μπορούμε να συνάψουμε αυτές τις συμφωνίες, τι γίνεται με αυτά τα σκάφη, θα επιστρέψουν στα ευρωπαϊκά ύδατα και ε, ως εκ τούτου θα ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στα αποθέματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε όλοι τη διακυβεύεται. Μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία και είναι προφανές ε, ε, ότι μπορούμε να συνάψουμε συμφωνίες στο μέτρο που ε, συμμορφώνονται με τους κανονισμούς περί παράνομης λαθρείας και αναρχής αλίας. Ε, όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν συναυθούν οι συμφωνίες θα ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στα δικά μας αποθέματα. Είναι αμφίδρομη η διαδικασία, δηλαδή και η, κράτη, τα κράτη, και Ευρωπαϊκή Ένωση που να κάνει προσπάθειες και τα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν σημαίες τρίτων χωρών και αλλιεύουν σε διαδικασία τα Μην ξεχνάτε ότι αυτό θα σημάνει μεγαλύτερη πίστα από θέματα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλα και ο κύριο Πένοστο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια μετά από τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις που έκανε η συναδελφή σα. Όντω, είναι κίτρινη κάρτα, κύριε Ρόμεβα. Πρέπει να πω όμω ότι η Επιτροπή δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να σταματήσει εδώ. Είπα ότι τόσο για αυτέ τι χώρε με την κίτρινη κάρτα. Θα αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία και θα δούμε αν θα σηκώσουμε κόκκινη κάρτα στο τέλο, αλλά θα δούμε ακριβώ τι κάνουν και όχι μόνο αυτέ οι μικρέ χώρε, αλλά άλλε Αυτές τις, αυτά τα δύο χρόνια Έχουμε επισκεφθεί και εμείς αυτά τα μεγάλα ψάρια, όπως είπατε, και θα συνεχίσουμε να τα επισκεφτόμαστε, τουλάχιστον κάποια από αυτά. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι κάποια από αυτά τα μεγάλα ψάρια, κάποιο από αυτά, το έχουμε επισκεφθεί και αντέδρασε θετικά. Πολύ. Διότι συνειδητοποίησε όχι μόνο τους κινδύνους της ε, εμπορίας ε, ε, των αλλιευμάτων αυτών, αλλά το τι σημαίνει αυτό για την φήμη του και παραέξω το ότι ακολουθεί τέτοιες πρακτικές. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός και θα πρέπει να δούμε επίσης γιατί κάποιες χώρες συμπεριλάβονται και γιατί κάποιες όχι. Τώρα, το θέμα λίστας με τα σκάφη μπαίνουμε σε ένα θέμα το οποίο εσά σα ενδιαφέρει πάρα πολύ και θέλετε να έχετε πολύ περισσότερε προφορίε. Αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συνεχίζει η Επιτροπή να εργάζεται για ενδεχόμενη ε, κατάλογο αλλιευτικών σκαφών που επιδίδονται στην παράνομη αλληλεία. Αλία. Για ποιο λόγο. Πολύ απλή εξήγηση και δεν έχει να κάνει τίποτε με έλλειψη πολιτικής βούλησης. Θα ήθελα να επιβληθώ τις ευκαιρίες για να σας πω ότι η Επιτροπή έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ε, πολιτική βούληση να εφαρμόσει τον κανονισμό κατά της παράνομης αλίας. Να μην έχετε καμία αμφιβολία. Ελέγχθη αυτό και από εμά και από την Κομισιόν και από την Επίτροπο. Θέλουμε όντως το θέμα αυτό να το πάμε μέχρι τέλους. Για ποιο λόγο καθυστερούμε, διότι πρόκειται για ένα νέο μέσον για ένα μέσο το οποίο η νομική ε, υπηρεσία θέλει να είναι από νομικής πλευράς απολύτως σίγουρη για το ότι θα γίνει και θα ήθελα να σας πω και κάτι από άποψη στρατηγικής. Όπως ξέρετε όλοι και συμφωνείτε, αυτός ο κανονισμός δεν είναι για να εφαρμόσουμε τώρα κάποια μέτρα και να το ξεχάσουμε. Πρόκειται για πολιτική μακροπρόθεσμη. Και σε αυτή την μακροπρόθεσμη πολιτική είναι θεμελιώδου σημασία να μην κάνουμε τίποτε το οποίο θα αποδυναμώσει την ε, ισχύ του νομικού πλαισίου στο οποίο θα κινούμεθα. Τι κάνουμε τώρα. Έχουμε σε ένα κατάλογο, θέλουμε να έχουμε ένα κατάλογο στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται ε, αμφιβόλου σοβαρότητας χώρες ή σκάφη, διότι αν μπούμε ε, σε αυτή την δυναμική και αρχίσουμε μετά από προσφυγές στο δικαστήριο να χάνουμε τις υποθέσεις, θα καταστραφεί ό,τι κάνουμε στα πλαίσια αυτού του κανονισμού για την εξάλληψη, εξάλληψη της παράνομης κλαθρίας και άναρχη αλίας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε τα βήματα που κάνουμε να είναι πάρα πολύ ισχυρά από νομική πλευράς, να μην μπορεί κανείς να μας προσβάλλει στα δικαστήρια όχι ότι δεν θα συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει να ελαχιστοποιήσουμε τις περιπτώσεις τις οποίες ενδεχομένως θα χάναμε σε δικαστήριο. Διότι αν αρχίσουμε μία μετά την άλλη σε όλες τις περιπτώσεις να έχουμε προσφυγές στα δικαστήρια και να χάνουμε, τα έχουμε χάσει όλα. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε, επαναλαμβάνω, για να έχουμε την νομική βεβαιότητα ότι ό,τι κάνουμε είναι σωστό και επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα νέο ε, μέσον, με ένα νέο εργαλείο νομικής προβλήσης για το οποίο δεν έχουμε και καμία νομολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη η νομική υπηρεσία θέλει να προχωρεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και γι' αυτό υπάρχουν καθυστερήσεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η απόφαση της Επιτροπής, εάν δείτε, είναι η πιο παράξενη στην δομή της από αυτές που έχω δει εγώ τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι έχει περισσότερες από 420 παραγράφους για δύο σειρές απόφαση, για δύο σειρές διατάφτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσες αποδείξεις και στοιχεία χρειάζεται για να σηκώσει κανείς την κίτρινη κάρτα. Και αυτό που συμβαίνει με τα λεφτικά σκάφη είναι ακριβώς το ίδιο. Γι' αυτό κύριε Ρωμέβα θα το λέω αυτό. Ασχολούμεθα με το θέμα αυτό Τώρα, πόσα λευτικά σκάφη θα συμπεριλάβουμε στον κατάλογο δεν ξέρω. Είμαστε εν μέσω τη διαδικασία. Αν καθυστερούμε και αν είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι διότι θέλουμε να έχουμε τη νομική εγγύηση και την νομική ασφάλεια την ε, μεγαλύτερη δυνατή. Ποτέ δεν είμαστε προστατευμένοι 100%. Εν περιπτώσει, τώρα να σα πω και ένα αστιάκι από αυτό που μα αφορά στην Κομισιό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σχέδιο κανονισμού στον οποίο υπάρχουν ε, τα, για τα αλληλεκτικά σκάφη και έχουμε ε, αιτιολογικές ε, σκέψεις και παραγράφεται ε, στην, στο συλλογιστικό περισσότερες από 800. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εσείς μπορεί να θεωρείτε ότι είναι απελπιστική η καθυστέρηση, αλλά εμείς σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Τώρα, σε σχέση με αυτό που για την αμφιστημία τη Κομισιόν, κυρία Φράγκα. Διαφωνώ, διότι όπω σα είπα ήδη, η Κομισιόν θέλει να πάει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο σε αυτό το θέμα. Και ίσως η διαδικασία της ε, ε, διαβούλευσης το 22 Οκτωβρίου δημιούργησε σύγχυση. Όντω υπάρχει σύγχυση. Η σύγχυση όμω δεν πρόκειται από το γεγονό ότι η Κομισιόν δεν έχει πολιτική βούλαση με πλήρη διαφάνεια, πρέπει να σας πω ότι όντως είδαμε ότι υπάρχει σφάλμα στον κανονισμό και ποτέ δεν ήταν του νομοθέτη η πρόσθεση ε, πριν να βγάλει κίτρινη κάρτα να βγάζει την κόκκινη με το καλημέρα σας. Όπως λέμε, πάντα θα πρέπει να σηκώνουμε από την κίτρινη κάρτα και μετά την κόκκινη. Ποιος είναι ο λόγος και από νομική που έγινε αυτή η σύγχυση που δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα διότι στη διαβούλευση 22 Οκτωβρίου είπε κάποια χώρα ότι λαμβάνοντας υπόψη τη διασταύρωση στοιχείων που προβλέπονται, η εφαρμογή αυτής της κίτρινης κάρτας σημαίνει ότι θα πρέπει αμέσως να εφαρμοστούν εμπορικές κυρώσεις. Και αυτό δεν ήταν ποτέ η πρόθεση του νομοθέτη. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν οι κατάλληλε διορθώσει ώστε να μην επαναληφθεί αυτό το πρόβλημα και στο μέλλον. Σα το αναγγέλλω λοιπόν αν δεν το έχετε. Ενημερωθεί, δεν έχετε ενημερωθεί μέχρι τώρα, ότι παρουσιάζουμε μια τροπημένη πρόταση, όχι για να αλλάξει η πολιτική μας, αλλά για να γίνει αυτή η, διευκρίνηση διευκρίνηση όσον αφορά την αρχική πρόθεση του νομοθέτη. Πρώτα σηκώνουμε την κίτρινη κάρτα και μετά την κόκκινη. Ε, δημιουργήθηκε το σφάλμα και σύγχυση διότι δεν ήταν σαφή τα πράγματα. Επίσης, Είπε η κυρία Φράγκο το άρθρο 31 ήδη είχε εφαρμοστεί στον Παναμά και σε άλλες χώρες. Όντω στον Παναμά και σε άλλες χώρες είχε γίνει προειδοποίηση, αλλά όχι επισήμω μέσω πράξη τη Επιτροπής. Οι αξιωματούχοι τη Επιτροπής είχαν, εμείς είχαμε ειδοποιήσει τον Παναμά και τις άλλες 8 χώρες ότι αν δεν βελτιώσουν ε, την κατάσταση και δεν επομισθούν τις ε, ε, ευθύνε του θα εφαρμοστεί ο κανονισμό περί παράνομη Αυτό έκανε, κυρία Φράγκα, πολλέ φορέ η Κομισιό. Προειδοποίησε τον Παναμά και άλλε χώρε για το τι συνέβαινε. Αλλά αυτό ανεπισήμω, ω προειδοποίηση, ω και ω επίσημη απόφαση της Επιτροπής. Την κυρία Λόβιν. Θα πω το εξή, ότι όντω λάβαμε υπόψη το γεγονός ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με κίτρινη χώρα για τις χώρες, αλλά μια σοβαρή προειδοποίηση και προς τους εφοπλιστές, τους Ευρωπαίους και όσους είναι πλειοκτήτες τέτοιου είδους αλλιευτικών σκαφών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν Ευρωπαίοι πλειοκτήτες που σκέφτονται «Πού θα πάω τώρα το σκάφος μου εγώ» και αυτό αφορά όχι μόνο τις χώρες που θα παω τωρα το σκαφος μου εγω και αυτο φορα οχι μονο τις ε, ε, αλλά και τους πλειοκτήτες και τους εφοπλιστές. Και τους λέμε ότι ακούστε, εάν ε, είμαι σε μία χώρα στην οποία γίνονται έλεγχοι και εγώ κάνω παράνομες πράγματα, ε, κάποια στιγμή θα με πιάσουν. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι εμείς προσπαθούμε να έχουμε ενισχυμένη συνεργασία και με κάποιες χώρες όπως είπα και η Ιαπωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ίσως ο μεγάλο περιορισμό τον οποίο έχει αυτός ο κανονισμός είναι ότι είναι μονομερής. Κανονισμός τη ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι έχουμε ε, ως κατάσταση. Βλέπουμε κάποια πλοία ε, τα οποία έχουν σημαία μία από τις χώρες ε, μία από τις χώρες τις οποίες εξετάζουμε που άλλαξαν σημαία. Εάν λοιπόν μακροπρόθεσμα δεν μπορέσουμε οι μεγάλες αλλιευτικές εμπορικές αγορές του κόσμου να συνεργαστούμε, αντί να λύσουμε το πρόβλημα το μεταθέτουμε, το μεταφέρουμε. Θα χρειαστεί ε, χρόνος, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή τον κύκλο που έχουμε αρχίσει να τον εξετάζουμε να τον κλείσουμε. Διότι ε, θα πρέπει οι χώρες ε, που ενεργούν παράνομα να ξέρουν ότι κάποια στιγμή τον αλλιευτικό του στόλο, τον οποίο εμεί ελέγχουμε, δεν θα μπορέσουν ε, κάποιοι να τον πουλήσουν ε, ούτε στη ΣΥΠΑ ούτε στην Ιαπωνία για να συνεχίζει να αλλιεύει με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε και στο μέλλον, ώστε να μπορέσουμε και στο μέλλον να έχουμε πολυμερή συνεργασία, την καλύτερη δυνατή. Και ε, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που αν επιτρέπετε θα αναφέρω και αφορά το θέμα των νομικών εγγύσεων. Ένα από τα θέματα για τα οποία θέλουν να είναι στην νομική μας υπηρεσία σίγουροι οι συνάδελφοι είναι ότι και σε επίπεδο κρατών και σε επίπεδο σκαφών δεν θα μπορεί κανείς εύκολα να κάνει προσφυγές κατά του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Ένα από τα καλύτερα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο ένωσης για να προστατεύσουμε το μέσον αυτό από τέτοιου είδους περιπτώσεις που προσφύγουν στον ΠΟΗ είναι κάθε φορά ό,τι κάνουμε να το κάνουμε όλο και πιο πολυμερές διότι μόνον έτσι θα μπορούμε να το προστατεύουμε και στο επίπεδο του ΠΟΕ. Είναι και θέμα στρατηγική αυτό και μεγάλη σημασία. Και συνεχίζουμε εδώ τι προσπάθειες. Η κυρία Λέβιν είπε ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τρία μεγάλα προβλήματα έχουμε προβλήματα τα οποία θα θέλουμε να επιλύσουν τα κράτη-μέλη. Τα προβλήματα που προέρχονται από την δυνατότητά τους να ελέγχουν τα σκάφη τους. Είναι πρωταρχική σημασία να υπάρχει σύστημα κυρώσεων. Κάποιες από αυτές τις χώρες δεν έχουν τέτοιο σύστημα επιβολής κυρώσεων. Και αν τα σκάφη τους, τα σκάφη με τη δική τους σημαία ε, πέφτουν σε σημαντικά παραπτώματα δεν ε, υφίστανται κυρώσει. διότι δεν υπάρχει σε κάποιε περιπτώσει ούτε καν και κείμενη νομοθεσία. Και όταν υπάρχει και εφαρμόζεται είναι ανεπαρκής. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε συστήματα κυρώσεων στι χώρε. Δεύτερον, θα πρέπει οι χώρε αυτέ να έχουν ένα ελάχιστο ε, σύστημα και, τα, και αυτό είναι απαραίτητο σε αναπτυσσόμενε χώρε, ένα ελάχιστο σύστημα ελέγχου των σκαφών του. Υπάρχουν κάποιε χώρε που δεν έχουν VMS και αν κάποιο πει ε, το τάδε σκάφος με δική σας σημαία μου λένε ότι ε, επιδίδεται σε παράνομη αλία στο τάδε μέρος. Αν μου πει κάποιος δεν μπορώ να παρακολουθήσω και την πορεία του σκάφους και δεν ξέρω πού βρίσκεται και τι κάνει, τι να κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό κάποιες χώρες και να μπορούν να εντοπίζουν ε, πού δραστηριοποιούνται τα σκάφη τους. Τώρα, σχέση με αυτό που είπε ο κ. Γκάλαχερ, νομίζω ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η κοινοτική ε, πλειοκτήτες και επιχειρηματίες τους οποίους ενδιαφέρουν ε, σκάφη με ξένες σημαίες να θέλουν να τα επαναπατρίσουν στα κοινοτικά ύδατα. Υπάρχουν μέτρα που το δυσκολεύουν, μην το κάνουν αυτό αδύνατο. Και δεύτερον, στην πράξη οι περισσότεροι ε, κοινοτικοί επιχειρηματίες και πλειοκτήτες που έχουν πλοία σε τέτοιες χώρες ε, έχουν σκάφη τα οποία ποτέ δεν αλίευσαν σε κοινοτικά ύδατα, κυρίως σε διεθνή ύδατα και σε ύδατα τρίτων χωρών. Γι' αυτό, εάν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για κάποιο σκάφος που αλλιεύει στα τροπικά ύδατα τόνο ή ε, αλλιεύει με παραγάδια, δεν νομίζω ότι θα έρθει στα δικά μας κοινωτικά ιδέα. Δεν λέω από την νομικής πλευρά αυτό είναι αδυνατό. Υπάρχουν όμως τόσο πολλά εμπόδια και αν δούμε ποιες δυσκολίες σημαίνει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος. Επίσης, εάν θέλουμε να, με την απαγόρευση τη ρητή, να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην αλλαγή της σημαίας των σκαφών, είμαστε υπέρ το να λάβουμε οποιοδήποτε συμπληρωματικό μέτρο χρειάζεται για να ενισχυθεί όλη αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πένας. Βλέπω ότι δεν ζητείτε ε, να, από κανέναν να λάβει το λόγο. Το επόμενο θέμα, όπως σας είχα αναγγείλει, είναι το θέμα της ανταλλαγής απόψεων μετά από τις ε, συνεδριάσεις που έγιναν στα πλαίσια της 18ης ε, συνάντησης της ΙΚΑΤ. Τι θέλετε να κάνουμε σήμερα το απόγευμα, περιμένουμε τώρα. Δύο-τρία μέλη μόνο είμαστε εδώ και δύο είμαστε παρόντες. Τι θέλετε, θέλετε να κάνουμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων, δεδομένου ότι τώρα έχουμε χρόνο. Ο κύριος Ρωμέβα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Το θέμα για μένα είναι αρκετά απλό. Διότι είχαμε την δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε ένα μέρος αυτής της συνάντησης. Η συνάντηση κράτησε δέκα μέρες. Κάποιες μέρες είμαστε παρόντες και η εντύπωσή μου δεδομένου ότι ήταν η τέταρτη συμμετοχή μου σε μια τέτοια συνάντηση της ΙΚΑΤ, είναι ότι σαφώς ε, για κάποια θέματα βλέπουμε αποτελέσματα. Καλό είναι αυτό και θα πρέπει να εξηγήσουμε και να πούμε ότι κάποια μέτρα όντως έχουν θετικές επιπτώσεις. Καλό είναι επίσης να εξηγήσουμε ότι όσον αφορά το θέμα ανάκτησης του ερυθρού τόνου, παρά το γεγονός ότι ακόμη είναι ανεπαρκή τα βήματα, οι επιστήμονες λέγουν ότι καλά τα κάνουμε τα πράγματα ενδεχομένως, αλλά μας ζητούν περισσότερο χρόνο για να το επαληθεύσουμε και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η ΚΑΤ για το θέμα αυτό είναι ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστό το αίτημα που υπέβαλε η Επιστημονική Επιτροπή. Νομίζω καλή απόφαση, άλλες φορές επικρίναμε τις αποφάσεις. Μια στιγμή Ραούλ περίμενε. Υπάρχει πάλι πρόβλημα ε, με την ε, διερμηνία στα γερμανικά. Όλα καλά. Έλεγα λοιπόν ότι όπως άλλες φορές κάναμε πάρα πολύ αυστηρές επικρίσεις ε, στην αποφάση κάτι που δεν έλαβε υπόψη τα, ε, την άποψη των επιστημόνων για το θέμα αυτό το ερυθρού τόνου, η σύσταση που έγινε να μην ξεπεραστούν τα, ε, οι 13.000 τόνοι, και αν λάβουμε υπόψη ότι η Αλγερία είχε ένα πρόβλημα από πέρσι, είμαστε σε... θα είμαστε δύο χρόνια σε μια ποσότητα ε, τάκ 13.500 τόνων. Επίσης, θέλω να πω ότι υπάρχουν ακόμη πολλές περιπτώσεις που δεν έχουν αποσαφινιστεί όσον αφορά κακές πρακτικές. Και αναφέρομαι και στην ε, παράνομη αλληλεία. Υπάρχουν κάποιες πρακτικές που κάποιοι δεν θέλησαν να εξετάσουν με τη σοβαρότητα τη δέουσα. Πιστεύω ότι για να είναι τέτοιου είδους οργανώσεις αξιόπιστες θα πρέπει τέτοιου είδους περιπτώσεις να εξετάζουν μεγάλη σοβαρότητα. Και θα πρέπει να μην επωφελούμεθα τις ευκαιρίες ε, να ε, καταγγέλλονται, αφού καταγγελθούν κάποιες περιπτώσεις, να γίνονται ιδέουσες έρευνες. Ας μιλήσω για τον Παναμά. Τώρα, αυτό εμάς μας ενδιαφέρει ως Ισπανούς πάρα πολύ. Υπάρχει το θέμα επίση των εισαγωγών τη Ιαπωνία, Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που θέλω να αναφέρω είναι κάτι το αρνητικό. Μπορούμε να πούμε ότι με αυτά τα οποία έγιναν ε, βελτιώθηκε η κατάσταση προς το παρόν για τον ερυθρότων, αλλά για τους καρχαρίες, τι να πω, όλα είναι αρνητικά. Ούτως ή άλλες, στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε με τρόπο σημαντικό. Εάν είχαμε ψηφίσει, όπως είναι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από την συνάντηση του ΙΚΑΤ, πάρα πολλά από τα προβλήματα που είχαμε στην ΙΚΑΤ δεν θα είχαν συμβεί. Μεταξύ άλλων, διότι η Επιτροπή στη συζήτηση που κάναμε για τα ε, ότι θα πρέπει οι καρχαρίες να εκφορτώνονται πριν ε, να semanas antes del voto en el Pleno, eh, evidentemente. τα περίγεια είναι κάτι που δεν θα μας είχε δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό που έγινε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σημαντικό, θα έπρεπε ίσως να το είχαμε κάνει στο παρελθόν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα πρέπει να το παραγνωρίσουμε. Και τελικά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην παραγνωρίσουμε την σημασία της διαρθρωτικής συζήτησης, στην ΕΚΑΤ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διαδικασία αναθεώρησης της ε, εντολής της ΕΚΑΤ, της ε, τρόπου λειτουργίας και νομίζω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, κάποια προβλήματα στην ΕΚΑΤ και τα οποία θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να διορθωθούν. Τα λέω όλα αυτά επιγραμματικά, γιατί ήταν τα βασικά κατά την άποψή μου. Ευχαριστώ κυρία Φράγκα. Κύριε... Ο κύριος Ρωμέβα από τη δική του άποψη εξήγησε κάποια πράγματα. Υπάρχουν ε, θέματα με τον οποίο την ερμηνεία συμφωνώ. Αλλά για κάποια θέματα πρέπει να υπάρχει και μία αιτιολόγηση. Το θέμα του ερυθρού ε, τόνου λύθηκε προς το παρόν. Και είδαμε ότι όπως πριν από δύο χρόνια, πριν να προτείνουμε πάρα πολύ εντυπωσιακά μέτρα, περιμένοντας είδαμε ότι τα πράγματα λειτουργούν και όλα αποδείχθηκαν ότι και όπως αποδείχθηκε ήταν πολύ καλό το σχέδιο που είχαμε υιοθετήσει και σήμερα η κατάσταση για τον ερυθρό ήταν καλύτερη από τον Βακαλάο. Πολύ σωστές αποφάσεις ελήφθηκαν και το 2014 θα γίνει επανεκτίμηση, διότι αν συνεχίζει να πηγαίνει καλά η κατάσταση για τον ερυθρό τόνο, τότε χώρες όπως το Μαρόκο, όπως είπαν, και αν είναι αρκετά καλά τα αποθέματα και δεν αυξηθούν τα τάκ, μπορούμε να οδηγηθούμε και σε παρανομή Θα είναι χειρότερη κατάσταση. Τώρα αναφορά τις τρεις προτάσεις για τους καρχαρίες, τη μία η ΕΠΑ και την ανέφερε ε, ε, ο κύριος Ρωμέβα και συνάδει με αυτά τα οποία ψηφίσαμε την άλλη φορά, πρέπει να πω ότι κανένας δεν την υποστήριξε. Η συζήτηση κράτησε δύο λεπτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε καν ε, άνοιξε στόμα της. Κανένας δεν συμφωνούσε με την πρόταση που έγινε και πρέπει να πω ότι χώρες όπως η Ταϊβάν που είναι από τις λίγες χώρες που απαγορεύει την ε, εκφόρτωση με αυτό τον τρόπο και είναι από τις λίγες χώρες που έχουν ε, ε, σκάφη κατάψυξης και απαγορεύει να εκφορτώνεται ο Καρχαρίας με ή χωρίς πτερήγια, Ε, δεν είπα τίποτε δεδομένου ότι όταν ε, ε, γίνει απόψυξη για να κοπούν τα πτερίγια μειώνεται η ποιότητα του αλλιεύματος. Τώρα, το κόστος για μας θα είναι πάρα πολύ υψηλό και αυτοί οι οποίοι αλλιεύουν σε ποστά 93% και εμεί σε 7% θα κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχουν χώρες τις οποίες πάντα θεωρούμε εξαιρετικά και συντηρητικά και ε, ε, που είναι για την διατήρηση των διαφόρων ειδών, όπως ο Καναδάς. Υπάρχει ένα ψάρι το οποίο απαγορεύεται να αλλιεύουμε εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Λάμια και αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του ε, Καρχαρία και πάλι. Δεν νομίζω ότι ενεργήσαμε σωστά. Θα έπρεπε ίσως να περιμένουμε την απόφαση της ΙΚΑΤ και μετά να πάρουμε εμείς αποφάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι τέτοιου είδους μέτρα λαμβάνονται και πολλές φορές πρέπει να γυρίσουν αντίον μας. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι δημοσίως εκφράζω την αντίθεσή μου και την δυσαρέσκεια μου, διότι ε, πάρα διότι πάρα πολλοί βουλευτές που ήθελαν να πάνε δεν μπόρεσαν να πάνε και πήγαν άλλοι που δεν κάνανε ίσως τίποτα. Το λέγω αυτό διότι όπως βλέπετε εδώ πέρα πιο πολλοί απόντες παρά παρόντες είμαστε και δεν καταλαβαίνετε πόσο κακό είναι αυτό όταν έχουμε μια την προσωπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά από τόσες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουμε να βλέπουμε ότι πήγαν κάποιοι και δεν εμφανίστηκαν και διότι δύο μέρες πριν είπαν ότι δεν θέλουν να πάνε. Δεν είναι σωστό αυτό, διότι χάνουν την ευκαιρία συνάδελφοι που θέλουν να πάνε και ενδιαφέρονται. Αυτό είναι έλλειψη συναδελφικότητα εκ μέρου συναδέλφων και θέλω να το πούμε κυρίω αυτού οι οποίοι πάντα είναι οι πρώτοι που βάζουν το όνομά του και δεν πάνε ποτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πάκα. Δεν έχω... Πα... Κάρμεν. Δεν έχω κι εγώ να προσθέσω πολλά πράγματα και εγώ κάποιε μέρε ήμουν παρόν και όντω Βλέπω ότι υπάρχουν δύο πάρα πολύ σαφείς ε, θέσεις που εκφράστηκαν. Όντες όμως το θέμα του Καρχαρία υπήρχαν πάρα πολύ σαφείς ε, θέσεις. Σε κάποιους άρεσαν, σε κάποιους δεν άρεσαν. Για τους λόγους που δεν θα αναφέρω, η θέση της Κομισιόν ήταν αυτή που είναι και όσον αφορά τον ε, κόκκινο τόνο. Βλέπουμε ότι τώρα τα πράγματα, τον ερυθρό με συγχωρείτε τα πράγματα είναι καλύτερα και είναι ευχάριστο αυτό. Τώρα, οι αποσίες είναι σοβαρό θέμα. Και πρέπει να σας πω ότι για μένα ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό. Διότι έκανα με την Προεδρία τρομερό αγώνα για να μας επιτρέψουν να πάμε. Δεν επέτρεψαν να πάμε έξι από την Επιτροπή μας, μόνο τρία άτομα. Ε, κινητοποιηθήκαμε σε όλες τις πολιτικές ομάδες, ανταλλάξαμε επιστολές, ε, στείλαμε επιστολές στη γραμματεία, στο Προεδρείο, στη Γενική Γραμματεία. γιατί επειδή είχαμε δίκιο, τελικά μας επέτρεψαν να πάμε έξι άτομα και εκτός εμού που είμαι εκτός ποσόστοσης, τελικά πήγαν δύο. Δύο και πρόεδρος. Πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, μας δημιουργεί πρόβλημα για το πώς μπορούμε σε τέτοιου είδους ε, διεθνείς συναντήσεις να έχουμε παρουσία και πώς ε, ε, έχουν τα πράγματα και ποια είναι η θέση μας σε σχέση με το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τρεις μόνο αντί για έξι συνεγώ είναι πολύ μέτριο. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Έχουμε γίνει σαν τους ιερείς στην εκκλησία που μιλάει στους παρόντες της λειτουργίας αλλά απευθύνεται με τον τρόπο αυτό και στους απόντες. Τι να κάνουμε τελικά. Πόσοι είμαστε εδώ και πόσοι κυρίως είμαστε παρόντες στις συνεδριάσεις πρέπει να δούμε. Ήταν εξαιρετικά τυχές που στο τέλος ε, δεν ε, ε, μπορούσαν να πάνε διάφορα μέλη της Επιτροπής και το ίδιο ισχύει με τον WCPFC. Ο κύριος Γκρόμπετς, η κυρία Φράγα και εσείς ο ίδιος δεν θα μπορέσετε τελικά να πάτε καταλαβαίνω ότι αποφασίστηκε το πράγμα τελευταία στιγμή, άλλαξαν γνώμη στη διάσκεψη των προέδρων και αυτό ήταν ατυχές και δημιούργησε τα προβλήματα. Ελπίζω αυτό να μην επηρεάσει ε, το ενδεχόμενο διοργάνωσης αποστολής ε, στο μέλλον, ε, διότι ήταν λάθος της διάσκεψης των Προέδρων που δεν μπόρεσαν όλοι να προγραμματίσουν εκ των προτέρων το ταξίδι ε, ίσως θα έπρεπε να το συζητήσουμε περαιτέρω πώς γίνεται η κατανομή ε, για τις αποστολές ούτως ώστε όλοι όσοι έχουν ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για το ζήτημα να έχουν τη δυνατότητα να πάνε πρόεδρος. Ε, ναι, προβλέπετε αύριο να το συζητήσουμε αυτό το θέμα για τις χειρεύουσες θέσεις, για τους αντικαταστάτες ε, σε σχέση με τις αποστολές. Οπότε θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Κυρία Ρόντουστ, ε, ναι, καταλαβαίνω αυτά που λέτε και... Αλλά ήθελα να κάνω μία πρόταση. Συνεχίζουμε και μιλάμε για ένα σωρό πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά πριν από την ψηφοφορία μια ανακοίνωση της Προεδρίας, όταν βρίσκονται όλοι οι βουλευτές εδώ στην αίθουσα, διότι δεν έχει νόημα να κάνουμε να κάνουμε προσκλήσεις. Πρέπει ουσιαστικά να κατηγορήσουμε αυτούς και οι ευθύνε ε, πρέπει να απευθύνουν στις πλάτες των πολιτικών ομάδων. Οι συντονιστές είναι εκείνοι που πρέπει να λένε ότι τα μέλη της εκαστή ομάδας ε, Οι συντονιστές υπάρχουν για αυτό το σκοπό, γι' αυτό υπάρχουν και συνεδρία των συντονιστών. Θα δούμε τι θα γίνει με τους συντονιστές και θα τα δούμε απευθείας ε, στην Ολομέλεια. Πάντως, ε, ο συντονιστής σε κάθε πολιτική ομάδα είναι εκείνος που πρέπει να μεριμνήσει ε, ώστε οι βουλευτές του να καταλάβουν τις επιπτώσεις κάθε απόφασης. Μόνο έτσι μπορούμε να δουλέψουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι το θέμα είναι ποιος θα υποφεληθεί 2, 3, 10. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι συντονιστές πρέπει στις πολιτικές πολιτικές ομάδες να καταβάλουν μια συγκεκριμένη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση γιατί είναι μικρή η Επιτροπή μας. Έχουμε 25 αναπληρωματικά μέλη ε, και ο μέσος όρος είναι 7, 8 ή 9 μέλη της ε, Επιτροπής, ε, οπότε πιστεύω ότι έχει σημασία όχι μόνο σε σχέση με αυτά που κάνουμε τώρα, αλλά και σε σχέση με τις μελλοντικέ εργασίε μας. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο και δεδομένων και των αλλαγών που έχουμε κάνει στην μερίσια διάταξη, θα ε, κηρύξω τη λήξη της, ε, συνεδρίασης, ε, της πρωινής συνεδρίασής μας. Θα είναι φορτωμένο το απόγευμά μας. Διακόπτουμε τώρα. Να όχι ένα λεπτάκι. Η Επιτροπή έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Silencio, por favor. Eh, no había dado la palabra a la Comisión en relación con ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που δίνετε και στην Κομισιόν την ευκαιρία να σας ενημερώσει κάπως ε, για τα αποτελέσματα της 16ης ε, συνεδρίασης της Διεθνούς Επιτρόπης ε, για την προστασία των θηνοειδών που έλαβε χώρα τον Νοεμβρίο στο Αγκαντήρ του Μαρόκο. Τα σημεία κλειδιά αναφέρθηκαν ήδη ε, από τους ευρωβουλευτές, ουσιαστικά ο ερυθρό Τόνος και οι Καρχαρίες κυρίως, αλλά θα προσπαθήσω να σας δώσω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τι συνέβη σε αυτή τη σύνοδο. Αυτό που ήταν καλό ήταν ότι η συμμετοχή ενδιαφερομένων ήταν η μεγαλύτερη από ποτέ. 41 από τα 48 μέρη ήταν παρόντα. Αυτό οφείλεται στη θετικά αποτελέσματα ε, της δημιουργίας ενός Ταμείου Ανάπτυξης ε, για τις αναπτυσσόμενες χώρες που καθιερώθηκε πέρυσι. Αλλά πρέπει να σας πω ότι και η συμμετοχή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν εντυπωσιακή. 100 άτομα αποτελούμενα από μέλη διοικήσεων κρατών μελών ε, του τομέα, περιφερειακά συμβούλια και επίσης και μέλη της Επιτροπής αυτής μας τίμησαν και φυσικά θα θέλαμε να ήταν εκεί και άλλα μέλη που είχαν ανακοινώσει ότι θα ήταν εκεί. Ελπίζω αυτό να συμβεί στην επόμενη σύνοδο. Θα σας προσώσω τα κύρια αποτελέσματα της συνόδου. Θα ξεκινήσω με τα μέτρα διατήρησης. Θα θυμάστε ότι στην τελευταία συνάντηση έγιναν πολλές συζητήσεις για διάφορα αποθέματα και υιοθετήθηκαν διάφορα μέτρα διατήρησης αποθεμάτων καθώς και μακροπρόθεσμα ε, σχέδια για τους μεσογειακούς ψηφίες και για τον ερθρό τόνο και φέτος εστιαστήκαμε σε νέα αποθέματα για τα οποία υπήρχαν νέες αξιολογήσεις, δηλαδή ερθρό τόνο και καρχαρίες. Ε, είναι πολύ σημαντικό ότι τόσο για, τον ερυθροτονό, για τα δύο αποθέματα τόνου, δυτικά και ανατολικά, δείξαμε ότι εξακολουθείται η υπεύθυνη προσέγγιση για τη διαχείριση των αλλιευμάτων. Και τα δύο αποθέματα ε, τέθηκαν σε επίπεδα που τηρούσαν τις, συμβουλές, τις επιστημονικές συμβουλές για τον ερθρό τόνο. Το ΤΑΚ ε, τέθηκε στους 13.400 ε, τόνους. Επίσης 100 ε, τόνοι δόθηκαν στην Αλγερία, αντιστάθμιση του τι έγινε το 2010. Συνολικά το επίπεδο συνολικών επιτροπόμενων αλλιευμάτων αναγνωρίζει ότι υπάρχει ανάκτηση των εχθείων ενώ ταυτόχρονα αυτό το επίπεδο ΤΑΚ μας επιτρέπει να είμαστε προσεκτικοί δεδομένοι στις ε, αβεβαίες ταχύτητες της ανάκτησης. Επίσης και πιστεύω αυτό είναι σημαντικό, η ε, μικρή αύξηση του ΤΑΚ αναγνωρίζει τις προσπάθειες των αλλιέων τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκτησης που θέτει ένα αυστηρό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Προβλέπεται ενημερωμένη αξιολόγηση για το 2014 του αποθέματος και θα τεθούν νέα μοντέλα το 2015. Επίσης είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τον ερυθρό τόνο τόσο στα δυτικά όσο και στα ανατολικά ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση και αναθεώρηση του πολιετούς σχεδίου ανάκτησης λαμβάνει υπόψη νέες εξελίξεις και προσπαθεί να απλουστεύσει ε, ε, τα μέτρα και αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή ICAT. Επίσης, το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του ρηθρού τόνου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις 16 Μαΐου του χρόνου με μια μεταβατική περίοδο για όσους δεν καταφέρουν να το υλοποιήσουν ένα πλήρως ε, σύστημα ηλεκτρονικό όσον αφορά τον ερθρό τόνο. Παρότι έγιναν κάποιες προσπάθειες αύξησης του ΤΑΚ ε, πέραν των ευλογονορίων, οι 15 τόνοι ε, που ισχύουν τώρα ε, θα ισχύσουν και για του χρόνου. Ταυτόχρονα μεταφέρονται του χρόνου και ταυτόχρονα υπάρχει ένα σχέδιο ανάκτησης για τον ερυθρό τόνο. τέθηκαν τα όρια σε 195.000 τόνους και 355.000 τόνους. Το μερίδιο είναι... Ε, έτσι θα επιτραπεί να ληφθούν υπόψη διάφοροι τρόποι που έχουμε αλλιεύσει στην Ευρωπαϊκή Τώρα τα μέτρα για τον ξηφία μεταφέρονται επειδή η αξιόλογηση θα λάβει χώρα του χρόνου. Για τους Καρχαρίες ε, τώρα, γιατί συζητήθηκε ήδη το θέμα, ε, ε, η πρόταση για περιορισμό των αλλιευμάτων στα τωρινά επίπεδα, όπως προτείνουν οι επιστημονικές συμβουλές για τη ζήγενα, αλλά και για άλλα είδη καρχαριών, τελικά δεν υποστηρίχθηκαν, αλλά έχουμε στο περιθώριο της συνεδρίασης διαπιστώσει τη δυνατότητα να συναυθεί συμφωνία με τον Καναδά ε, μετά από συζητήσεις για τα συμβαλόμενα μέρη ε, καταλήξαμε στο ότι δύσκολα θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε μια εξαίρεση για τον ε, Καναδά αλλά άρα ούτε και για άλλα συμβαλόμενα μέρη. Σε σχέση τώρα με τα πτερίγια που διπλώνονται πάνω στο σώμα του Καρχαρία δεν πέρασε η πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αν μπορούσε και, να μπορούσε μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει το λόγο και να υποστηρίξει αυτή την πρόταση, θα είχαν αντιταχθεί οι ασιατικέ χώρε. Αυτό οπότε δεν θα περνούσε η πρόταση για του καραχαρίε, Πάντω, η πρόταση για να βελτιώσουμε την συμμόρφωση με τα ισχύοντα μέτρα για του Καραχαρίε, υποστηρίχθηκε Οπότε εν γέννη λυπούμεθα που η ΆΙΚΑΤ αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει για την προστασία των καρχαριών ε, για διάφορους λόγους όπως το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης ΆΙΚΑΤ και από αυτή την πλευρά είναι πολύ καλά τα νέα ε, της ε, τροποποίησης, της απόφασης τροποποίησης της σύμβασης ΆΙΚΑΤ από πλευρά της ΆΙΚΑΤ για συγκεκριμένα στη σημεία όπως παραδείγματος χάρη καρχαρίες, μακροπρόθεσμη προστασία των καρχαριών αλλά και βελτιώσεις σε άλλους τομείς για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας, παραδείγματος χάρη διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ο ρόλος των μη συμβαλωμένων μερών της σύμβασης. Ε, κατά αυτά για τα αποθέματα, τώρα θα ήθελα να σχολιάσω άλλα ζητήματα που δεν σχετίζονται με τα αποθέματα, αλλά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία επίσης. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος ε, για το καθεστώς ε, διαχείρισης ε, και ελέγχου που είναι εφαρμοστέο στην ICAT. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελάχιστα πρότυπα για τον έλεγχο στους λιμένες εγκρίθηκε και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή των, της συμφωνίας για τα μέτρα ελέγχου των κρατών λιμένα σε σχέση τώρα με το καθεστώς τεκμηρίωση των αλλιευμάτων για άλλα είδη θηνοειδών ο ερυθρός τόνος ξεκίνησε και είχαμε και αναθεώρηση του Γενικού Μέτρου για τις τα φορτώσεις, εξασφαλίζοντας έτσι ε, τις εμπλό μεταμορφώσεις, καλύτερο έλεγχο δηλαδή για τις εμπλό μεταφορτώσεις, ε, σε σχέση με το EBCD τώρα και τον ερυθρό τόνο ε, η ΆΙΚΑΤ κατάφερε με αυτά τα μέτρα να ενισχύσει την ικανότητά της φέτος να καταπολεμεί την παράνομη άναρχη και λαθρέα αλία. Εν γέννη βελτιώθηκε η συμμόρφωση με τους, κανόνε με, τους κανόνες ε, ΆΙΚΑΤ από πλευράς των συμβαλωμένων μερών, δηλαδή βελτιώνονται τα αποτελέσματα ε, και δεν είχαμε μόνο από πλευράς πέντε συμβαλωμένων μερών ε, ε, επιστολές ταυτοποίησης προβλημάτων. Το, τα αποτελέσματα από την περσινή χρονιά ήταν καλή σε σχέση με την πιστοποίηση BCD και την εγκυρότητα κάποιων επιστημονικών στοιχείων. Αναμένουμε ακόμη τα στοιχεία, αλλά ούτως ή άλλως πρόκειται για την πρώτη όχληση που μπορεί να λάβει ένα συμβαλόμενο μέρος και μπορεί να μην φτάσουμε καν σε επιστολή σχολείο που καταγράφει ουσιαστική ανησυχία και δεν είναι μια απλή ειδοποίηση. Ε, έχει περάσει και ο χρόνος τώρα. Ε, νομίζω, για να συνοψίζω σιγά σιγά, ότι στην επόμενη ετήσια συνέλευση ε, της ΑΕΚΑΤ στο Cape στην Νότιο Αφρική στις 16 με 26 Δεκεμβρίου ε, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αποτελεσματικά τις θέσεις μας. Σας ευχαριστούμε. Υπάρχει κανένας που θα ήθελε το λόγο. Όχι, διακοπή λοιπόν τη συνεδρίαση μέχρι τις 3 όπου θα καταφτάσει ο Επίτροπος Δεγκούχτ.